Good afternoon. Bonjour. Buenas tardes. Everybody take a seat. Ready to go. Καλησπέρα. Καθίστε παρακαλώ για να ξεκινήσουμε. Please be welcome to this session. Καλώς ήρθατε σε αυτή τη συνεδρία της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ. Το πρώτο σημείο, ως συνήθως, concerns the το πρώτο σημείο αφορά την έγκριση της ημερήσιας διάταξης, ο συνήθως. Σας προτείνω λοιπόν να εγκρίνουμε το σχέδιο ημερήσιας διάταξης με κάποιες μικρές αλλαγές. Πρώτον, το σημείο 3 και το σημείο 7 να τα συζητήσουμε μαζί. Έχουν σχέση με, τη, με το μέλλον της συνθήκης της Λισαβόνας. Το 3 θα το συζητήσουμε λοιπόν μαζί με το 7. Μετά θα γίνει η ανταλλαγή απόψεων με τον, με τον ε, εισηγητή μας για το σύστημα αξιολόγηση Schengen που αφορά και την θέση ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας. Και σημειώστε ότι τις ίδιες αυτές εκθέσεις θα τις ψηφίσουμε αύριο το πρωί. Και μετά στις 5 θα συζητήσουμε με τον συντονιστή για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, τον κύριο Ζίλντα Κέρχοφ. Είναι ένα σημαντικό σημείο της ημερήσιας διάταξης για σήμερα. Αύριο θα παρακολουθήσουμε την ημερήσια διάταξη όπως έχει στο σχέδιο, εκτός από το σημείο 23 για τη μεταφορά των διαδικασιών σε ποινικέ υποθέσεις που μεταφέρεται στις 15 Οκτωβρίου, στην επόμενη συνεδρίαση. Υπάρχουν αντιρρήσεις μήπως? Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσει, εγκρίνεται η ημερήσια διάταξη. Περνάμε στο επόμενο σημείο, σημείο 2, ανακοινώσεις του Προέδρου. Δεν έχω καμία άλλη ανακοίνωση, παρά μόνο ότι μπορούμε να εορτάσουμε το δεύτερο δημοψήφισμα της Ιρλανδίας, που μας έφερε όλους πιο κοντά στο να δούμε τη θέση σε ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας ε, μέχρι τα τέλη του έτους ή αρχές του 2010. Φαντάζομαι ότι είναι καλά νέα αυτά για όλους μας. Και το σημείο 3 αφορά τον αντίκτυπο της συνθήκης της Λισαβόνας στο χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Στόχος αυτής της ανταλλαγής απόψεων είναι να ακούσουμε την νομική υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τη Σουηδική Προεδρία, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον εισηγητή της Επιτροπής ΑΦΚΟ που θα μας μιλήσουν για τη συνθήκη της Λισαβόνας. Ευχαριστώ την προσοχή σας στα βασικά σημεία του αντικτύπου της συνθήκης της Λισαβόνας στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Πρώτον, θα κρατήσουμε την συνεργασία Σέγγεν ως ε, κατευθυντήρια δύναμη του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Δεύτερον, οι πολιτικές στρέφονται από τη συνεργασία δημοσίων διοικήσεων στην προστασία θεμελιωδών δικαιωμάτων. Τρίτον, θα δώσει μεγαλύτερες δυνατότητες στους πολίτες της Ευρώπης που είναι η βάση της νομιμοποίησης του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα θα τηρούν την αρχή της ισότητας μεταξύ των πολιτών οι οποίοι θα την χάνουν ίσης προσοχής από τα κοινοτικά θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της κοινότητας. Τέταρτον, θα γίνει πιο αξιόπιστη η δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί θα βασίζεται σε μια νέα νομική βάση. Πέμπτον, θα απλουστεύσει το θεσμικό πλαίσιο καταργώντας την τρέχουσα διάσταση μεταξύ του πρώτου πυλώνα και του διακυβερνητικής, διακυβερνητικής πτυχής με τον τρίτο πυλώνα που δημιουργήθηκε από την συνθήκη του Μάστριχτ. Έκτον, θα ενισχύσει τη διαδικασία λήψη αποφάσεων και θα, έχει, θα δώσει μεγαλύτερε δυνατότητε στην ειδική πλειοψηφία στο Συμβούλιο. Έβδομον, θα βασίζονται στην αρχή της επικουρικότητας και της αναλογικότητας πολλά στοιχεία στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Και τέλος, ε, θα ενισχύσει τις δημοκρατικές αρχές με την ενίσχυση της συναπόφασης, διαδικασίας συναπόφασης μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλων αρχών λήψης απόφασης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα δώσω τώρα το λόγο καταρχήν στην νομική υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο κύριος Μπράντλεϊ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η σύντομη παρουσίασή μου σήμερα είναι συμπληρωματική προς τη δική σας παρουσίαση που ήταν ευσύνοπτη και πληρέστατη πολιτική ανάλυση. Εγώ θα δώσω μια περισσότερο θεσμική και νομική ανάλυση. Κύριε Πρόεδρε, η συνθήκη της Λισαβόνας θα ολοκληρώσει μια διαδικασία που ξεκίνησε με τη συνθήκη του Μάστριχ το 1993 για να εφαρμοστεί η κοινοτική μέθοδος της κατάρτισης και εφαρμογής πολιτικών στον χώρο της ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Η νέα συνθήκη που απλουστεύει σημαντικά και εκδημοκρατικοποιεί την λήψη αποφάσεων σε αυτό τον τομέα και λέω απλουστεύει διότι θα υπάρχει μια ε, νομική διαδικασία η οποία θα ισχύει παντού η κανονική, η απλή νομική διαδικασία που είναι το νέο όνομα για τη ε, διαδικασία της συναπόφασης. Και τα Εθνικά Κοινοβούλια και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έχουν σημαντικό ρόλο στην έγκριση και εφαρμογή των μέτρων αυτών. Το θεσμικό πλαίσιο στο χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης θα κρατήσει κάποια βασικά γνωρίσματα, αλλά αυτά θα είναι περιορισμένα και στο μέλλον. Η ε, απλή νομοθετική διαδικασία θα ισχύει σε όλους τους τομείς ε, συμπεριλαμβανομένων και των ε, τομέων όπου τώρα δεν συμπεριλαμβάνεται η διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπω είναι οι διεθνεί συμφωνίε. Θα θυμάστε τη συμφωνία SWIFT που συζήτησε τον περασμένο μήνα η Επιτροπή, τη συμφωνία SWIFT με τι Ηνωμένες Πολιτείες. Θέματα τα οποία συζητούνταν υπό τον τρίτο πυλώνα, όπω η δικαστική συνεργασία σε ποινικέ υποθέσει και η αστυνομική συνεργασία, το εξή θα συζητώνται με τους ίδιους κανόνες που ισχύουν για την εσωτερική αγορά αυτή τη στιγμή τα μέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών σε αυτούς τους ε, τομείς ε, θα υπόκεινται σε νομική εξέταση από το ε, Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Τίθενται λοιπόν νέοι στόχοι από τη Συνθήκη της Λισαβόνας για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει ως απέτηση η αλληλεγγύη μεταξύ κρατών μελών, ώστε να είναι δίκαια και προς πολίτες τρίτων χωρών. Και εδώ οι συνιστώσεις είναι το άσυλο και ο έλεγχος στα εξωτερικά σύνορα, όπως επίσης και οι στόχοι της διευκόλυνσης τη των πολιτών στη δικαιοσύνη. Υπάρχουν δύο συγκεκριμένα θεσμικά γνωρίσματα που ισχύουν οριζόντια σε όλους τους τομείς ασφάλεια ελευθερίας και δικαιοσύνης. Το πρώτο είναι ότι τα εθνικά κοινοβούλια θα παίζουν ένα πιο έντονο ρόλο και για την έγκριση μέτρων με την εφαρμογή των πρωτοκόλων για την ε, επικουρικότητα και για τον κανονισμό των Εθνικών Κοινοβουλίων και στο χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης υπάρχει μια ιδιαιτερότητα όσον αφορά την αξιολόγηση της εφαρμογής αυτών των πολιτικών συμπεριλαμβανομένης και της συνεργασία για την ασφάλεια και τι δραστηριότητε της Eurojust και της Europol. Το δεύτερο γνώρισμα, και αυτό δεν είναι τίποτα καινούριο, είναι ότι η Δανία, η Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο εποφελούνται ε, από ένα ειδικό καθεστώς opt-out ε, με βάση τα σχετικά πρωτόκολλα στι συνθήκε. Επίσης υπάρχουν και κάποια συγκεκριμένα γνωρίσματα τη συνθήκη της Λισαβόνας που περιορίζονται σε συγκεκριμένε αποφάσεις ή κατηγορίες αποφάσεων και όχι σε πλήρης τομείς κατάρτισης πολιτικής σχετικά με τα άτομα προς τα οποία ε, και είναι περιορισμένα ω προς τα άτομα στα οποία εφαρμόζονται ή ε, σε σχέση με τι χρονικέ περιόδου κατά τι οποίε ε, εφαρμόζονται. Ένα τέτοιο στοιχείο είναι η διαβούλευση με το Κοινοβούλιο σε τομεί όπω ε, μέτρα προσωρινή συνεργασία όταν αντιμετωπίζουμε μαζική εισρωή υπηκόνων τρίτων κρατών ή οικογενειακά ζητήματα, θέματα οικογενειακού ε, δικαίου που εμπλέκουν ε, διεθνή συνεργασία ή αστυνομικέ δράσει από αστυνομική δύναμη μια χώρα σε επικράτη άλλου κράτου μέλου. Κάποια από αυτά τα μέτρα απαιτούν ομοφωνία στο Συμβούλιο και απλή διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και όχι την, ειδική, την ψήφιση με ειδική πλειοψηφία. Τρίτον, όσον αφορά την νομική συνεργασία σε ποινικέ υποθέσει και αστυνομική συνεργασία, η Επιτροπή θα πρέπει να έχει το δικαίωμα πρωτοβουλία από κοινού και με άλλου. Οκτώ κράτη-μέλη προς το παρόν δεν διέπονται από, αυτή την, από αυτόν τον κανόνα. Και ε, επίσης υπάρχει δυνατότητα να εφαρμόζουν τα κράτη-μέλη ε, μια, μια διακοπή επίγουσας ανάγκη σε θέματα αστυνομική συνεργασίας και δικαστικής συνεργασίας όταν επηρεάζονται ε, τα, συστήματα, τα δικαστικά συστήματα των κρατών μελών. Το σχέδιο νομική πράξη ε, θα ψηφίζεται με συνένεση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και αν δεν μπορεί να επιτευχθεί συνένεση, τα κράτη-μέλη που θέλουν να προχωρήσουν θα μπορέσουν να εφαρμόζουν την ενισχυμένη συνεργασία. Το τελευταίο ειδικό γνώρισμα που θα ήθελα να αναφέρω περιορίζεται και ω προ το χρόνο και ω προ το πεδίο εφαρμογή και αφορά νομικέ πράξει τη Ευρωπαϊκή Ένωση που αφορούν την αστυνομική συνεργασία, δικαστική συνεργασία σε ποινικέ υποθέσει και εγκρίνονται σύμφωνα με το καθεστώ που ισχύει πριν από τη Λισαβόνα. Για μια πενταετή περίοδο μετά τη θέση ισχύ τη συνθήκη τη Λισαβόνα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα μπορεί να ε, ξεκινά διαδικασίε επί παραβάση για κράτη-μέλη που δεν εφαρμόζουν αυτά τα μέτρα και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θα μπορεί να, θα μπορεί να δίνει προδικαστικά... Ε, ε, απαντήσει σε προδικαστικά ερωτήματα σύμφωνα με το περιορισμένο καθεστώ το οποίο ήδη εφαρμόζεται. Κύριε Πρόεδρε, ασχολήθηκα με τι εξαιρέσει στους κανόνες. Θα πρέπει να είναι σαφές ότι ο γενικός κανόνας το εξή θα είναι ότι η κατάρτιση πολιτικής στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης ε, είναι κοινοτικοποιημένο απολύτω τώρα πια, εκτό από αυτέ τι εξαιρέσει που ανέφερα. Ε, μία από τι βασικέ επιπτώσει τη θέση σε ισχύ που θα ήθελα να αναφέρω είναι ότι ο χάρτη των ανθρωπίνων των θεμελιωδών δικαιωμάτων θα έχει την ίδια νομική αξία όπω και οι συνθήκε τα κράτη, τα, οι ευρωβουλευτέ ε, σίγουρα είναι εξοικειωμένοι με τις εγγύσει των θεμελιωδών δικαιωμάτων που ισχύουν ε, και γνωρίζουν ότι προστατεύονται τα θεμελιώδη δικαιώματα από την κοινοτική νομική τάξη και αυτά θα επεκτείνονται και στο δεύτερο και στον τρίτο πυλώνα. Θέλω όμω να τονίσω άλλη μια φορά τα όρια, δηλαδή αντί να περιγράψω το πεδίο εφαρμογή, θα περιγράψω τι εξαιρεσει που υπάρχουν. Καταρχήν ο χάρτης θεμελιωδών δικαιωμάτων είναι σαφέ ότι δεν επεκτείνει τι ε, αρμοδιότητε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, όπω ορίζονται στις συνθήκε. Δηλαδή το πρώτο που θα πρέπει να εξετάσουμε είναι το εύρο τη νομοθετική δυνατότητα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, όπω προκύπτει από τη νομική βάση τη συνθήκη. Ο Χάρτη. Ε, θα επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο ασκούνται αυτές οι αρμοδιότητες και ε, όσον αφορά τα θεσμικά όργανα και όσον αφορά ε, τα όρια των εξουσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και θα σας δώσω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Ε, κανόνες για την προστασία των δεδομένων που υιοθετούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη το άρθρο 8 και τις απαιτήσεις του άρθρου 8 του χάρτη. Δηλαδή ότι όλοι έχουν δικαίωμα προστασίας των προσωπικών τους δεδομένων δίκαιη επεξεργασία για συγκεκριμένους στόχους επιτρέπεται, αλλά μόνο επί τη βάση συνένεσης ή ε, κάποια άλλη νομική βάση που θα θεσπίζεται δια νόμου. Και τρίτον, ε, οι κοινοτικοί οι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει ε, να εξασφαλίζουν ότι κάποια ανεξάρτητη αρχή διαβεβαιώνει τη συμμόρφωση προς τους κανόνες. Τα δικαιώματα με βάση το χάρτη διατυπώνονται στα άρθρα από 1 49, αλλά το άρθρο 52 ε, δηλώνει ότι η άσκησή τους μπορεί να περιορίζεται και πάλι εξαίρεση της εξαίρεσης μπορούν να περιορίζονται μόνο σύμφωνα με ε, το δίκαιο, σύμφωνα ε, με την τήρηση της διεθνούς τάξης όταν είναι, υποχρε... όταν είναι απαραίτητος ο περιορισμός αυτών των δικαιωμάτων και όταν υπάρχουν σαφώς πραγματικοί στόχοι συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ή ανάγκη προστασίας δικαιωμάτων άλλων. Όσον αφορά το πεδίο της προσωπικής εφαρμογής, ο χάρτης είναι απολύτως δεσμευτικός προς όλα τα θεσμικά όργανα, όλους τους οργανισμούς και όλες τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλες τις δραστηριότητές τους. Επίσης δεσμεύει τα κράτη-μέλη, αλλά μόνο όταν εφαρμόζουν δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ε, και υπάρχει κάποιο ειδικό πρωτόκολλο για το Ηνωμένο Βασίλειο και την Πολωνία. Τελευταίο σημείο που θα ήθελα να αναφέρω αφορά την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και το αποτελεί αρμοδιότητα και υποχρέωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, που θα πρέπει να προσυπογράψει το χάρτη των, των θεμελιωδών δικαιωμάτων και εδώ υπάρχει στο άρθρο 6 παράγραφος 2 της νέας συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, μέχρι τώρα να προσχωρήσει σε αυτή τη συνθήκη. Μετά την συνθήκη τη Λισαβόνα θα μπορέσει να διαπραγματευτεί την ένταξη, την προσχώρηση η Επιτροπή και το Συμβούλιο θα πρέπει να ε, υπογράψει τι απαραίτητε συμφωνίε. και θα πρέπει να υπάρξει και συνένεση του, Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και έγκριση από τα κράτη-μέλη σύμφωνα με τι συνταγματικέ ε, διατάξει κάθε κράτου μέλους. Η προστιθέμενη αξία από αυτή τη διαδικασία είναι ότι θα υπάρχει μια διαδικασία μεμονωμένη άσκηση άσκησης ε, καταγγελίας ε, αλλά βέβαια η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορεί πάντοτε να παρέχει πιο ε, επεκταμένη συνεργασία από ό,τι στη σύμβαση μέχρι τώρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και αν υπάρχουν ερωτήσεις θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε είτε εγώ είτε οι συνάδελφοι. Now... Σας ευχαριστώ. Κύριε Περίλο, θέλετε να πείτε κάτι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δύο μικρές παρατηρήσεις να προσθέσω σε αυτά τα οποία είπε ο κύριος Μπράγκλη όσον αφορά την ένταξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Και τώρα επιτρέψτε μου να συνεχίσω στα γαλλικά. Οι συνθήκε τη Λισαβόνα πραγματικά προβλέπουν ε, ε, ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση να προσχωρήσει στη Σύμβαση για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πρώτα λοιπόν για υποχρέωση. Αλλά στη σύμβαση που μιλά για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφέρεται ότι η διαδικασία αυτή προσχώρησης θα γίνει με βάση την, θα γίνει βάση ομοφωνία στο Συμβούλιο και θα ακολουθεί εθνική διαδικασία έγκρισης που σε, ε, σε γενικέ γραμμέ αντιστοιχεί ε, στη διαδικασία κύρωση, αλλά ευτυχώ η διαδικασία τη Λισαβόνα, ε, η συνθήκη τη Λισαβόνα δεν αναφέρεται στη διαδικασία με το όνομα κύρωση. Είναι σημαντικό η επιτροπή σα να επιμείνει στο εξή. Το άνοιγμα τη διαδικασία τη ένταξη τη Ευρωπαϊκή Ένωση στην Σύμβαση Ανθρώπινα Δικαιώματα να γίνει όσο το πιο γρήγορα και με όσο το πιο αποτελεσματικό τρόπο διότι η ένταξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα θα οδηγήσει σε μια κατάσταση που θα έχουμε ένα εξωτερικό έλεγχο, δηλαδή από το δικαστήριο του Στρασβούργου που ε, ο έλεγχος ασκείται σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θα υπάρξει κανένα κράτο το οποίο μπορεί να επιλέξει opt-out, πράγμα που προβλέπεται για, το χάρ, για τη Χάρτα των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Η ένταξη λοιπόν σύμβαση για τα ανθρώπινα δικαιώματα θα ανοίξει ακόμα περισσότερο τη ε, ε, διαδικασία τη Στοκχόλμη. Γιατί πάνω από τα 50% των σημείων της διαδικασίας και του προγράμματος Στοκχόλμης επηρεάζονται άμεσα από την ένταξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Λοιπόν, τώρα πάω στη δεύτερη πτυχή. Ότι πρόκειται για υποχρέωση είναι και άποψη του Δικαστηρίου της Γερμανίας ε, στην, στην απόφαση της 36ου του 2009. Το Συνταγματικό Δικαστήριο της Γερμανίας αναφέρεται και αυτό σε υποχρέωση ένταξης, προσχώρησης. Και το υπενθυμίζω εδώ διότι σε αυτή την απόφαση του δικαστηρίου της Καρσρούης υπάρχουν μακροσκελείς ε, ε, αναφορές στον Ευρωπαϊκό Δικαστικό Χώρο και κυρίως στην δικαστική ε, συνεργασία σε ποινικέ υποθέσεις. Όπως θα θυμάστε, σε αυτή την υπόθεση το Γερμανικό Δικαστήριο θεωρεί ότι ε, στο συγκεκριμένο θέμα, οι εκπρόσωποι τη ε, γερμανική κυβέρνηση, πριν, πριν πάρουν θέση στο Συμβούλιο, θα πρέπει να έχουν λάβει οδηγίε από την Ομοσπονδιακή Γερμανική Βουλή. Ε, αυτή ε, η απόφαση επικρίθηκε ιδιαίτερα αυστηρά από τότε που εκδόθηκε, αλλά θα ήθελα να πω το εξή. Όσον αφορά εμά, πιστεύω ότι το γεγονό ότι σε ποινικέ υποθέσει, ένα ποινικό ζήτημα, το δικαστήριο τη Καρσούη υπενθυμίζει ότι τα κοινοβούλια πρέπει πρώτα απ' όλα να παίρνουν θέση μα οδηγεί στο συμπέρασμα ότι και όσον αφορά το κοινοτικό ε, επίπεδο, το ευρωπαϊκό επίπεδο, βεβαίω προβλέπεται διαδικασία συναπόφαση, αλλά η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν θα πρέπει να είναι ε, κατωτέρου επίπεδου από τη θέση του ε, Κοινοβουλίου του Βερολίνου. Σε περίπτωση λοιπόν δικαστικής, ποινική δικαστικής συνεργασίας θα πρέπει να λαμβάνονται πολύ περισσότερο υπόψη και αυτό είναι μια περισσότερο πολιτική εξήγηση παρά νομική εξήγηση τη απόφαση του Δικαστηρίου τη Καρσούη, θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τι θέσει του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ε, θα μπορούσα να επανέλθω στην απόφαση, αν το επιθυμείτε, σε μια άλλη συνεδρίαση. Αλλά ήθελα να σα υπογραμμίσω αυτή την πτυχή. Ευχαριστώ. Thank Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Περίλο. Ίσως ε, η Σουηδική Προεδρία θέλει να πει κάτι. Σας παρακαλώ. Κύριος Νίλσον. Thank uh, Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αρχίζω λέγοντάς σας ότι αισθάνομαι και εγώ την ίδια ικανοποίηση με εσά για το αποτέλεσμα της προφορίας την περασμένη Παρασκευή στο Δουβλίνο. Η Σουηδική Προεδρία αισθάνεται πλήρη ικανοποίηση με την τελική έκβαση του δημοψηφίσματος, όπου το, το ναι επικράτησε τόσο μεγάλο ποσοστό. Να σα υπενθυμίσω βεβαίω ότι δεν ολοκληρώθηκε η διαδικασία. Ε, Κρεμούν ακόμα ορισμένε κυρώσει. Αλλά έχουμε υψηλέ προσδοκίε ότι όλα αυτά θα λυθούν στο όχι και το σαπότερο μέλλον. Επίση, πιστεύουμε ότι μπορούμε να πούμε ότι συμφωνούμε σε μεγάλο βαθμό με την ε, άποψή σας για την συνθήκη. Με αυτόν τον τρόπο η Ένωση θα γίνει και πιο ανοιχτή και πιο δημοκρατική αλλά και πιο αποτελεσματική. Όσον αφορά τη συναπόφαση και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, από ό,τι έμαθα, από 40 θα γίνουν 80 οι τομείς πολιτικής και σε αυτούς τους 80 τομείς Ε, θα έχουμε ξεπεράσει πλέον το δημοκρατικό έλλειμμα που είχε παρουσιαστεί ε, με τις προηγούμενες συνθήκες. Όσον αφορά τώρα την εφαρμογή της συνθήκης Λισαβόνας, ε, συνεχίζονται βεβαίως συζητήσεις. Κάθε προεδρία πρέπει να προετοιμάζεται και βεβαίω και στο συγκεκριμένο θέμα συνεχίζονται συζητήσει και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γιατί είναι πολλά τα σημεία τα οποία είναι σημαντικά και για μας και για σας. Και πιστεύω ότι αυτές οι συζητήσεις ε, εξελίσσονται ομαλά και θα ενημερωθείτε για τα αποτελέσματα συζητήσεων αυτών. Ε, φαντάζομαι και σε εσωτερικό επίπεδο θα ενημερωθείτε. Κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι αυτό που ήδη αναφέρθηκε είναι πρόκειται για το ζήτημα των θεμελιωδών δικαιωμάτων, θέμα το οποίο μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Ένα άλλο ζήτημα είναι τι θα γίνει με τη νομική, με την, με νομική βάση που θα αλλάξει με τη νέα συνθήκη. Εδώ εκφράζω την ευχή να ακολουθήσουμε το παράδειγμα της διαδικασίας που ακολουθήσαμε και όταν πήγαμε από το Μάστριχτ στο Άμστερνταμ. Δηλαδή, στενή συνεργασία της Προεδρίας και των εισηγητών για να καταλήξουμε σε ικανοποιητικά αποτελέσματα και για το Συμβούλιο και για το Κοινοβούλιο. Αυτό αφορά και τις αποφάσεις πλαίσιο, αλλά ε, και τις νομικές βάσεις σε πολλούς άλλους τομείς. Και σας διαβεβαιώνω, και το ξέρετε κι εσείς, ότι οι πρόεδροι μας είναι σε στενή επαφή με όλους τους συγητές που έχετε διορίσει στα διάφορα θέματα. Τέλος, να αναφερθώ σε ένα ζήτημα το οποίο μόλις αναφέρθηκε από το μέλος του Κοινοβουλίου ότι στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για Αναφέρομαι στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα ανθρώπινα δικαιώματα ήθελε, ε, αναφέρθηκε στην όσο το πιο γρήγορη προσχώρηση. Συμφωνώ απόλυτα. Και πιστεύω ότι αυτό ε, θα αποτελέσει βασικό χαρακτηριστικό της πρότασης που θα υποβληθεί για το πρόγραμμα της Στοκχόλμης σε ε, δύο εβδομάδες περίπου. Θα θέλαμε λοιπόν να ολοκληρωθούν οι διαδικασίε ώστε να πιο γρήγορα και με ώστε να τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. ευχαριστώ. Ευχαριστώ εκ μέρου ε, τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η κυρία Λάουρα Κοράδο. Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα ε, και η Επιτροπή χαίρεται ιδιαίτερα με την έκβαση του Ιρλανδικού δημοψηφίσματος και εμείς πιστεύουμε ότι οι διαδικασίε κύρωσης θα έχουν ολοκληρωθεί σύντομα από όλα τα κράτη-μέλη. όπω είπε και ο εκπρόσωπος της Προεδρίας. Και ε, καλωσορίζουμε τις καινοτομίες της συνθήκης της Λισαβόνας, μόλις αρχίσει να ισχύει και ιδιαίτερα τι ενισχυμένε αρμοδιότητε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τη διεύρυνση της συναπόφαση ε, στα περισσότερα ζητήματα ε, του, ε, του τομέα δικαιοσύνη και εσωτερικών υποθέσεων, όπω είπαν και οι νομικές υπηρεσίες, καθώς επίσης και στον με τον ενισχυμένο ρόλο των Εθνικών Κοινοβουλίων. Όπω είπε και ο πρόεδρο έχουν συνεχίζονται οι προετοιμασίε από μεριά Συμβουλίου και σε επίπεδο επιτροπή συνεχίζονται οι στο μέτρο βεβαίω των αρμοδιοτήτων μα και ιδιαίτερα όσον αφορά την προετοιμασία για την προσχώρηση τη Ευρωπαϊκή Ένωση στη Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, καθώ και σε άλλα ζητήματα που ήδη αναφέρθηκε, καθώ και σε άλλα ζητήματα που τώρα θα αποκτήσουν νέα νομική βάση με τη νέα συνθήκη, όπω για παράδειγμα η πρωτοβουλία των πολιτών κτλ. Όσον αφορά την αλλαγή της νομικής βάσης πολλών μέσων που εκκρεμούν αυτή τη στιγμή, όπως είπε και η Προεδρία, και εμείς ελπίζουμε να συνεργαστούμε ιδιαίτερα στενά μαζί σας στις διάφορες προτάσεις και ιδιαίτερα και με τους εισηγητές των διαφόρων προτάσεων έτσι ώστε να συνεχίσει η εργασία με επικοδομητικό τρόπο, ιδιαίτερα όσον αφορά τις προτάσεις αυτές που θα μετακινηθούν από τη διαβούλευση στην συναπόφαση. Για αυτές τις προτάσεις, όπως και στο παρελθόν, όταν, κάνα, όταν ε, ε, ε, ε πήγαμε από το Μάστριχ στο Άμστερνταμ, η Επιτροπή πριν από τη θέση ισχύ της νέας συνθήκης έκανε μια ανακοίνωση όμνιμπους που κάλυπτε προτάσεις από διάφορους τομείς πολιτικής, εκεί όπου έπρεπε να αλλάξει νομική βάση και πρότεινε και την τυπική τροπολογία ε, των προτάσεων ως προς την νομική βάση. Όσον αφορά τώρα τι προτάσεις του τρίτου πυλώνα, εδώ μιλάμε για διαφορετικής φύσεως πράξη. Εμείς βλέπουμε το θέμα ως εξή. Έτσι ερμηνεύουμε την αλλαγή της συνθήκης και την αλλαγή της νομική βάσης. Ότι αυτές οι προτάσεις ε, δεν θα ισχύουν πλέον ε, με την θέση σε ισχύ της συνθήκης και θα πρέπει να ε, υποβληθούν εκ νέου ως προτάσεις. Άρα το πρόβλημα είναι αν δεν έχουν εγκριθεί επίσημα μέχρι τη θέση σε ισχύ της συνθήκης. Και το σκεφτόμαστε λοιπόν και αυτό το πρόβλημα και ε, σκέφτομαι τι θα, σκεφτόμαστε τι θα γίνει με τις προτάσεις ε, με, βάση, με τη νέα βάση και αυτό αφορά όχι μόνο τις προτάσεις που εκκρεμούν, που δεν θα έχουν εγκριθεί όταν θα αρχίσει να ισχύει η νέα συνθήκη, αλλά και το υφιστάμενο και εκτιμένο στον τρίτο πυλώνα. Και εδώ εξετάζουμε τις πιθανές αλλαγές των παλαιών πράξεων τρίτου πυλώνα. Συνεχίζεται λοιπόν ο προβληματισμός και ε, οι πολιτικές προτεραιότητες βεβαίως θα πρέπει να οριστούν και από τη νέα Επιτροπή και ιδιαίτερα από τους νέους επιτρόπους που θα είναι υπεύθυνοι ε, για ε, το χαρτοφυλάκιο δικαιοσύνης εξωτερικών υποθέσεων. Θα θέλαμε λοιπόν ε, τη συμβολή του Κοινοβουλίου και τις προτάσεις σας για τις προτεραιότητες σε θέματα πολιτικής και όπως σας είπα είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε και να συζητήσουμε μαζί σας το όλο θέμα. Ευχαριστώ. Thank you. Now we... Ευχαριστώ. Θα ανοίξει λοιπόν η συζήτηση, να πάρουν τον λόγο όσοι το ζήτησαν. Ναι. Ρούιτα Ταβάρες παρακαλώ. I'm sorry, President, but I don't think I... Δεν νομίζω ότι ζήτησα τον λόγο. Ε, ε, κάνατε μάλλον κάποιο λάθος, κύριε Πρόεδρε. Ε, εν πάση περιπτώσει, σας ευχαριστώ όμως. Α, ο κύριος Ρωμαίος, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Έχουμε μια συγκεκριμένη ερώτηση όσον αφορά την χάρτα και το πρωτόκολλο σχετικά με το Ηνωμένο Βασίλειο και την Πολωνία. Θα μπορούσατε, σας παρακαλώ, να γίνετε πιο συγκεκριμένος λέγοντάς μας ποιες θα είναι οι συγκεκριμένες επιπτώσεις. Δηλαδή, ε, θα ληφθούν υπόψη ε, στις δύο περιπτώσεις οι γεωγραφικές, ας πούμε, συντεταγμένες ή τα πολιτικά στοιχεία ε, και να μας δώσετε συγκεκριμένα στοιχεία επ' αυτών. Ευχαριστώ, κυρία Λάτφορντ. Και η ερώτηση δική μου αφορά το πρωτόκολλο. Εάν κατάλαβα καλά, ή μάλλον να το θέσω διαφορετικά. Ο κύριος Bradley αναφέρθηκε ε, σε ένα μάλλον σκοτεινό ή ομιχλώδες πρωτόκολλο για το Ηνωμένο Βασίλειο και την ε, Πολωνία η ε, αντίληψή μου είναι διαφορετική με την έννοια ότι δεν έχω καταλάβει τι θα γίνει με το πρωτόκολλο και ποια θα είναι η επίπτωση. Ο κύριος Μπράντλι βεβαίως, ε, ε, από ό,τι κατάλαβα, είχε γραπτό κείμενο που καλό θα ήταν να το έχουμε και εμείς. Από την άλλη πλευρά όμως, η νομική υπηρεσία θα έπρεπε να μας δώσει και την άποψή της όσον αφορά το πρωτόκολλο. Αυτό θα ήταν πραγματικά εξαιρετικά ενδιαφέρον και θα ήθελα να ακούσω ε, και την απάντηση που θα δοθεί στην ερώτηση του κυρίου ε, ε, Ρομέβα. Επίσης, εάν κατάλαβα καλά αυτά που είπε ο συνάδελφος του κυρίου Μπράντλη, δηλαδή εάν και εφόσον η Ένωση προσχωρήσει στη συνθήκη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα υπάρξει εξωτερικός έλεγχος που θα αφορά όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν θα υπάρχει δυνατότητα opting out. Επομένω, εδώ διαφαίνεται το ενδιαφέρον σενάριο. Όποιος ε, αποκλειστεί από το πρωτόκολλο της Πολωνίας του Ηνωμένου Βασιλείου και δεν θα καλύπτεται λοιπόν από την χάρτα, παρόλα αυτά μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο του Στρασβούργου και να παραπονεθεί για τον τρόπο με τον οποίο το Ηνωμένο Βασίλειο ή η Πολωνία ε, ε, ε, καλύπτει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από ένα πρωτόκολλο που δεν εφαρμόζει. Δηλαδή θα υπάρξουν κάποιοι στο Ηνωμένο Βασίλειο που ενδεχομένως θα το εκμεταλλευτούν Μήπως θα μπορούσαμε να έχουμε και τη διαφορετική άποψη των, της νομικής υπηρεσίας, γιατί Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι θεωρούσαν ότι ενδεχομένως απομονώνονται από, κάποια, από, την, ε, ε, από την χάρτα. Τελικά βλέπουμε, διαπιστώνουμε ότι δεν απομονώνονται, δεν προστατεύονται κατά κάποιο τρόπο από τον δάκτυλο της δικαιοσύνης ε, και του δικαστηρίου του Στρασβούργου. Τελειώσατε? Ναι, ωραία, ωραία λέει ο Πρόεδρος, πάρα πολύ ωραία. Εξεπλάγεται γιατί δεν μακρηγόρησα. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Μπουζούτιλ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ, όπως και προηγούμενοι ομιλητές, να πω ότι με μεγάλη χαρά ακούσαμε την έκβαση του Ιρλανδικού Δημοψηφίσματος και ελπίζουμε βεβαίως ότι και η διαδικασία κύρωσης θα ολοκληρωθεί το ταχύτερο δυνατό και θα αρχίσει να θα σε ισχύ η συνθήκη. Θα ήθελα όμως να κάνω μια ευρύτερη σκέψη, κύριε Πρόεδρε, σχετικά με το τι μας διδάσκει η κατάσταση στην Ιρλανδία. Όπως και οι συνάδελφοι γνωρίζουν, ένα από τα κύρια μελήματα των Ιρλανδών ψηφοφόρων είχε να κάνει με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία έχει μια τάση να χώνεται πολύ στα εσωτερικά και την εθνική ζωή, την οικογενειακή ζωή των πολιτών της. Ε, πράγμα δηλαδή που ξεπερνάει τα όρια που θεωρούν αποδεκτά οι πολίτες. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να ζητήσω να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί σε οτιδήποτε κάνουμε σε αυτό το θεσμικό όργανο και τον τρόπο με τον οποίο το κάνουμε. Υπάρχει το οικογενειακό δίκαιο βεβαίω. Και είναι γεγονό ότι στην περίπτωση της Ιρλανδίας ε, προβληματίστηκαν πολλοί Ιρλανδοί σχετικά με το βαθμό στον οποίο ε, θα μπορούσε η Ευρωπαϊκή Ένωση να αλλάξει το δικό του αρχές. Όταν, αρχίσει, όταν τεθεί σε ισχύ λοιπόν είναι να επεμβει στις δικες τους αρχες οταν αρχισει οταν σε ισχυ λοιπον η συνθηκη της Λισαβόνας, πράγμα που ελπίζω ότι θα γίνει γρηγορότερα παρά αργότερα, θα πρέπει να προσέξουμε και να δείξουμε προσοχή, σύνεση, ε, αλλά και ε, να προστατεύσουμε τους πολίτες μας. Δεύτερον, θα πρέπει να δούμε λίγο τον τρόπο λειτουργίας της δικιάς μας Επιτροπής, κύριε Πρόεδρε, ε, διότι το νομοθετικό βάρος της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης των τομέων αυτών δηλαδή θα αυξηθεί οπωσδήποτε και επομένως η οργάνωση της εργασίας μας θα πρέπει να αντικατοπτρίζει το άχθος αυτό και θα πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι ε, θα δώσουμε τον κατάλληλο χρόνο ε, κυρίως στα νομοθετικά ε, θέματα γιατί αυτά είναι τα οποία θα αυξηθούν περισσότερο και που θα έχουν μεγαλύτερο αντίκτυπο στην εργασία μας. Επομένως θα πρέπει να προσέξουμε και την κατάρτιση της ημερησίας διάταξής μας. Ε, θα πρέπει να δούμε λοιπόν με ποιο τρόπο αυτό το νομοθετικό βάρος, ε, κύριε Πρόεδρε, ε, θα αντικατοπτριστεί κατά κάποιο τρόπο στην καθημερινή μας εργασία. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Χάουτεγκερ παρακαλώ. Eh, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, θα ήθελα και εγώ ε, καταρχάς να αξιολογήσω πάρα πολύ θετικά ε, την έκβαση τη, του δημοψηφίσματος της Ιρλανδίας την Παρασκευή. Μερικές φορές στην πολιτική μπορεί κανείς να είναι αισιόδοξο, αλλά και εξαιρετικά απογοητευμένος. Αλλά καταλαβαίνουμε ότι σε αυτή την περίπτωση αν το το αποτέλεσμα δεν ήταν θετικό, ε, θα βρισκόμαστε πραγματικά σε απόγνωση. Τώρα όμως είμαστε πιο αισιόδοξοι. Τώρα, μία παρατήρηση σχετικά του τι θα σημαίνει για μας και στον, για τον τομέα με τον οποίο ασχολούμαστε η συνθήκη της Λισαβόνα με την προϋπόθεση βεβαίω ότι θα τεθεί σε εφαρμογή γρήγορα. Το δυναμικό της ε, συνθήκης της ε, Λισαβόνας ε, για τον χώρο ελευθερίας και δικαιοσύνης δεν θα είναι δυνατόν να εφαρμοστεί εάν τα κράτη-μέλη δεν δείξουν παράλληλα και γενεοδορία όσον αφορά την παραχώρηση της ε, κυριαρχίας τους ή ενός τμήματος της ε, κυριαρχίας τους. Ε, μιλήσαμε πολύ για τη δικαστική συνεργασία, μιλήσαμε για συνεργασία σε ποινικέ υποθέσεις κτλ. Αλλά τίποτα δεν θα μπορέσει να υλοποιηθεί πραγματικά εάν δεν δείξουν γενεοδορία οι χώρες μέλη και ε, πρέπει να πω ότι το Συμβούλιο έχει μεγάλη δυσκολία στο να οικοδομήσει κοινά έγγραφα ε, γιατί είναι πολλά αυτά που πρέπει να οικοδομηθούν στην Ευρώπη και πολλά αυτά τα οποία θα πρέπει να γίνουν έτσι ώστε να δοθεί πνοή στη Λισαβόνα. Ξέρετε ότι ε, το πρώτο εξάμεινο του επόμενου έτους ε, θα αναλάβουμε εμείς την Προεδρία στο Συμβούλιο. Κοίτα, εγώ εργάζομαι μαζί με άλλους ε, συναδέλφους από άλλες πολιτικές ομάδες στην Ισπανία για την επεξεργασία μια συνένεση ανάμεσα στις πολιτικές ομάδες στην Ισπανία, στήριξη της Ισπανικής Προεδρίας. Λοιπόν, θέλω να ενημερώσω τους συναδέλφους εδώ στο Κοινοβούλιο ότι από ό,τι φαίνεται όλες οι πολιτικές ομάδες στην Ισπανία ήδη έχουμε συμφωνήσει να ζητήσουμε από την κυβέρνηση η θεμελιώδης προτεραιότητα της Προεδρίας μας στο θέμα αυτό να είναι ακριβώς το θέμα της κύρωσης ε, της, ε, του Ευρωπαϊκού Χάρτη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και ακριβώ ε, αυτό θα αποτελέσει μία από τι προτεραιότητε ε, ε, που θα θέσει η Προεδρία, η Ισπανική Προεδρία για το επόμενο εξάμεινο. Η κύρωση, το ξαναλέω. Αν είναι δυνατόν στο πρώτο εξάμεινο, αν όχι μέσα στο πρώτο χρόνο, μέσα στο χρόνο αυτό, η κύρωση. Γιατί οπως είπε και καποιος συναδελφος είναι θεμελιωδες το θέμα αυτό. Και από όλε τι απόψει. Και κάτι άλλο, η άλλη πρόταση προ την οποία εργαζόμαστε, αναφέρω πάντα στι προτεραιότητε είναι η επεξεργασία μιας οδηγίας ή ενός κανονισμού που θα αναπτύσσει ε, την, ε, αυτή την ε, νομοθετική δυνατότητα των πολιτών. Αυτό που θα επιτρέψει δηλαδή σε ένα εκατομμύριο πολίτες με τις υπογραφές τους να μπορέσουν να ξεκινήσουν αυτό που πολλέ φορέ ζητάμε και εμεί στο Κοινοβούλιο και θεωρούμε ότι λείπει. Περισσότερη πρωτοβουλία στο νομοθετικό τομέα. Μαζί με την έκθεση ε, ε τη προηγούμενη ε, ε, Επιτροπή ΑΦΚΟ, η Ισπανική Προεδρία θεωρεί ω μία από τι προτεραιότητε τη ακριβώς την περαιτέρω ανάπτυξη αυτής της νομοθετικής πρωτοβουλίας που θα ε, δώσει το δικαίωμα ε, ε, νομοθετικής πρωτοβουλίας στους πολίτες. Σας ευχαριστώ κυρία Ιντβελτ. Ευχαριστώ, Άκουσα όλους αυτούς ε, που εξέφρασαν τη χαρά τους για το αποτέλεσμα του Ιρλανδικού δημοψηφίσματος. Συμφωνώ και εγώ. Ήταν πολύ καλά τα αποτελέσματα. Ήταν ένα σίγουρο ναι. Δεν ήταν ένα ναι που μόλις τα κατάφερε. Ήταν ένα πολύ στεναρό ναι. Και έχω κάποιες γενικές παρατηρήσεις. Κάποιος, δεν θυμάμαι ποιος μιλητής, είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα θα μπορεί να ασχοληθεί με ένα νέο πεδίο δραστηριοτήτων και αυτό θα ήθελα να το εκφράσω κάπως καλύτερα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη είναι δραστηρία σε πολλούς τομείς πολιτικής, ιδιαίτερα στους τομείς με τους οποίους ασχολείται η Επιτροπή μας, αλλά όχι με τρόπο ιδιαίτερα δημοκρατικό και διαφανή. Και νομίζω ότι αυτό είναι το μεγάλο όφελος για τους πολίτες της Ευρώπης, ότι αυτές οι πολιτικές τώρα θα ανοιχτούν προς τα έξω και θα, συζητούνται, θα συζητούνται ανοιχτά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και συνεχίζοντας την ίδια γραμμή θα ήθελα να πω ότι τα σχόλια του συναδέλφου, του ιδιαίτερα αγαπητού συναδέλφου Σάιμον Μπουζουτήλ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, εμφανίζεται ως ε, ε, παρισφρίουσα στην προσωπική και οικογενειακή ζωή των πολιτών θα έλεγα ότι δεν ανακατευόμαστε καθόλου, προστατεύουμε την ιδιωτική ζωή των πολιτών και αυτοί που ανακατεύονται στις ζωές των πολιτών είναι οι εθνικές κυβερνήσεις ε, και ε, κάποιες ε, οργανώσεις που ανακατεύονται στη ζωή των πολιτών. Μια άλλη παρατήρηση τώρα. Χάρηκα με αυτό το οποίο ανέφερε η νομική υπηρεσία του Συμβουλίου για την απόφαση του Γερμανικού Συνταγματικού Δικαστηρίου της Καρσρούης. Διότι ανησυχώ για τις επιπτώσεις που θα μπορούσε να έχει. λέει κάποια ιδιαίτερα σημαντικά θέματα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Λέει ότι ποτέ δεν μπορεί να είναι πραγματικό κοινοβούλιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να εκπροσωπεί του πολίτε τη Ευρώπη για διάφορου λόγου. Ότι δεν έχουμε πραγματική αντιπολίτευση, δεν έχουμε πραγματική κυβέρνηση. Και βασικά διότι δεν είμαστε σαν το Γερμανικό Κοινοβούλιο. Αυτό λέει. Και αν το διαβάσετε προσεκτικά, διαβάσετε προσεκτικά αυτή την απόφαση, φαίνεται σαν να βάζει από την πίσω πόρτα ένα νέο δικαίωμα αρνησικυρία για τα εθνικά κοινοβούλια. Και θα ήθελα να ζητήσω από την Επιτροπή μα και από εσά, κύριε Πρόεδρε, αν είναι δυνατόν να έχουμε μία νομική αξιολόγηση από την νομική υπηρεσία του Συμβουλίου για τι πιθανέ επιπτώσει ε, τη απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου τη Καρλσρούη. Και μια τελευταία παρατήρηση, απαντώντα στα ευγενικά σχόλια του εκπροσώπου του Συμβουλίου. Χαίρομαι που άκουσα ότι το Συμβούλιο έχει την πρόθεση να συνεργάζεται στενά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, διότι ειλικρινά τη συνεργασία μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου μέχρι τώρα, εγώ δεν θα την έλεγα ιδιαίτερα συνεργάσιμη. Και είπατε ότι ήρθατε σε επαφές με τους ε, εισηγητές για όλα τα σχετικά θέματα. Να σας πω, εγώ είμαι εισηγήτρια για τη Europol και για τα προσωπικά δεδομένα και για το άνοιγμα των ε, εμπιστευτικών εγγράφων προς ε, τρίτους και δεν ήρθε κανεί σε επαφή μαζί μου από το Συμβούλιο και ήμουν ε, εισηγήτρια και για το πρόγραμμα για τα στοιχεία επιβατών, το PNR και το Κοινοβούλιο ζήτησε από το Συμβούλιο να συμμορφωθεί με τα αποτελέσματα του ψηφίσματο μα από τον Νοέμβριο πέρυσι και τώρα σχεδόν έχουμε φτάσει στο πρώτο έτος, την πρώτη επέτειο από τότε που είχαμε εκείνο το ψήφισμα πέρυσι τον Νοέμβριο και δεν έχω δει καμία απάντηση από το Συμβούλιο. Ελπίζω λοιπόν ριζικά να βελτιωθεί η κατάσταση της συνεργασίας με το Συμβούλιο και ιδιαίτερα μετά την έγκριση τη συνθήκη της Λισαβόνα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Ινβελ, το κύριος Άλμπρεχτ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να προσθέσω κι εγώ ένα παράδειγμα με μια ερώτηση προς τη Σουηδική Προεδρία. Γιατί βλέπουμε ότι μετά το δημοψήφισμα της Ιρλανδίας πρόκειται να εγκριθεί η συνθήκη της Λισαβόνας και θα ήθελα να ακούσω τι πιστεύει η Σουηδική Προεδρία για το επιχείρημα ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τώρα θα πρέπει ε, να συμφωνεί με, ε, το, με την κάλυψη του πεδίου ε, του τρίτου πυλώνα. Μήπως αυτό σημαίνει ότι θα έπρεπε να σκεφτούν την αναβολή της συμφωνίας SWIFT που είχαμε τον περασμένο μήνα, γιατί η Επιτροπή μας δυσκολεύτηκε πάρα πολύ να εξηγήσει γιατί δεν θέλουμε αυτή τη συμφωνία τώρα. Θα με ενδιέφερε η θέση της Σουηδικής Προεδρίας από αυτού. Ευχαριστώ. Ο κύριος Άλβαρο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα προσθέσω κι εγώ σε αυτό που είπε η συνάδελφος η Σόφη, ότι δεν είχαμε και τόσο θετικές εμπειρίες με το Συμβούλιο. Βέβαια πρέπει να πω ότι για το ε, θέμα που ήμουν εγώ εισηγητή ε, για τη συνεργασία στα Τελωνία όντως ήρθα σε επαφή μαζί μου από την Προεδρία του Συμβουλίου και αρκετά νωρί μάλιστα. Και σε σχέση με αυτό που είπε ο κ. Άλμπρεκτ ε, εγώ θα ήθελα να δω τι γίνεται με διάφορα νομικά θέματα με τα οποία εμείς δεν έχουμε ασχοληθεί καθόλου. Ίσως να μην το κατάλαβα καλά αλλά υπάρχουν άλλα θέματα. Υπάρχει η Συμφωνία SWIFT, το θέμα των πληροφοριών των στοιχείων επιβατών που είπε η Σόφη, το PNR και κάτι ακόμη. Αν δεν υπάρχει συμφωνία SWIFT πριν από την έγκριση της συνθήκης της Λισαβόνας, τι θα κάνουν οι αρχέ τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα πάνε στι αρχέ των ΗΠΑ και θα πούνε ότι τώρα θα τα ξανακάνουμε όλα από την αρχή, γιατί πρέπει τώρα να συμφωνήσει και το Συμβούλιο, ή θα το κάνουμε με δεύτερο πυλώνα, γιατί είναι θέμα εξωτερική πολιτική. Δεν θα έχουμε συναπόφαση σε αυτό. Θα αλλάξει η νομική βάση απομακρυνόμενοι από εμά ή προσεγγίζοντά μα. Αυτό είναι ένα από τα ζητήματα με του συνεχιζόμενου φακέλου, τα συνεχιζόμενα θέματα. Επίση, τα συνεχιζόμενα θέματα που δεν έχουν εγκριθεί επισήμω, που δεν έχουν δημοσιευθεί δηλαδή στην επίσημη εφημερίδα των κοινοτήτων, θα πρέπει να ξαναρχίσουν από την αρχή. Θα με ενδιαφέρε ίσω η διαδικασία Omnibus σε αυτή την περίπτωση, να δω πώ λειτουργεί. Γιατί όταν εγκρίθηκε το κοινοβούλιο, εγώ τότε τελείωνα το σχολείο, άρα δεν είμαι τόσο παλιό για να τα ξέρω ακριβώ. θα γίνει μια γενική τροποποίηση που θα λέει αλλάζει η νομική βάση ή θα αρχίσει κάποιος τριμερής διάλογος από την αρχή. Ε, είναι πολύ ενδιαφέρον το τι θα γίνει και είναι, πολλές, ε, είναι πολλά αυτά τα οποία θα πρέπει να γίνουν. Ε, σε σχέση με αυτά που μας είπε η νομική υπηρεσία θα ήθελα να πω ότι είναι πολλά φιλοσοφικής υφής ερωτήματα βλέπουμε καταρχήν με όλη αυτή τη διαδικασία πώ μπορεί μια χώρα να τραβήξει χειρόφρενο στη διαδικασία τη ενοποίηση. Αν η Μεγάλη Βρετανία μπορεί να τραβήξει χειρόφρενο σε ένα θέμα ενό πρωτοκόλου, παραδείγματο χάρη. Υπάρχει κάποιο νομικό όριο ή μπορεί μια χώρα που έχει κάποια πρωτόκολλα που την αποκλείουν από κάποιου τομεί πολιτική μπορεί να πει ναι, δεν συμπεριλαμβανόμαστε, δεν μα αρέσει και το σταματάμε τώρα. Μπορεί να είναι κάτι που βολεύει την εθνική πολιτική μια χώρα. Ποιο ξέρει. Θα ήταν ενδιαφέρον λοιπόν να ξέρουμε την απάντηση. Και επίση κάτι που θα μπορούσαν ίσω να συζητήσουν οι συντονιστέ αύριο ή να το σκεφτεί η Γραμματεία. Ήδη αναφέρθηκε ότι είναι τεράστια η δουλειά που έχουμε να κάνουμε και στην περασμένη θητεία τα τελευταία χρόνια είχαμε πάνω από 400 θέματα που πέρασαν από την Επιτροπή μα. Και δεν ξέρω πόσα θα έχουμε όταν θα έχουμε συναπόφαση. Ω μέλο τη Επιτροπή Προπολογισμού είδα ότι έχουμε αύξηση των δαπανών για προσωπικό του Κοινοβουλίου η Επιτροπή μας θα έχει δικαίωμα σε μεγαλύτερο αριθμό προσωπικού γιατί κάνουν καταπληκτική δουλειά όλοι αλλά δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα ε, γιατί θα έχουμε τον ίδιο αριθμό προσωπικού με τεράστια αύξηση του όγκου δουλειάς μας. Θα ήταν ενδιαφέρον λοιπόν να ξέρουμε αν ε, μπορεί να γίνει κάτι και να το συζητήσουν οι συντονιστές και να το λάβει υπόψη η γραμματεία. Ευχαριστώ. Κύριος Μπρόνς. Ευχαριστώ. Δεν θέλω να καταστρέψω εγώ την εορταστική ατμόσφαιρα για τα αποτελέσματα του Ιρλανδικού δημοψηφίσματο, κάθε άλλο. Αλλά οι Βρετανοί συντηρητικοί είπαν ότι θα προσπαθήσουν να επαναδιαπραγματευθούν κάποια σημεία τη συνθήκη Λισαβόνα που δεν είναι σαφή. Ε, αυτό ε, θα μπορέσει να γίνει με βάση τα αποτελέσματα των Βρετανικών εκλογών. Ευχαριστώ πολύ για τη σαφήνειά σας. Και θα ακούσουμε τώρα την απάντηση της νομικής υπηρεσίας. Uh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν ξέρω αν μπορώ να ικανοποιήσω τα ερωτήματα όλων των βουλευτών. Ε, σίγουρα αυτό που μπορώ να σας ε, ικανοποιήσω ω αίτημα είναι ότι θα σας δώσω το γραπτό μου κείμενο για να μπορέσετε να το διαβάσετε. Για το πρωτόκολλο δεν υπάρχει κάποια ε, νομική θέση, αλλά αν θέλει η Επιτροπή σα κάποια γραπτή νομική θέση, θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε στα ερωτήματα αυτά. Για το αν ισχύει σε συγκεκριμένα άτομα ή σε δικαστήρια, θα προσπαθήσουμε να το διευκρινίσουμε. Όσον αφορά το οικογενειακό δίκαιο, ο κ. Βουσουτήλ έχει δίκιο. Είναι ένα βασικό θέμα από αυτά που συζητήθηκαν στην Ιρλανδία και ένα από τα συνθήματα που χρησιμοποιήθηκαν ε, ήταν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα σας αφήνει να μοιράσετε το αγρόκτημά σας. Αλλά από ξέρω δεν υπάρχει αρμοδιότητα Ευρωπαϊκής Ένωσης για οικογενειακά ζητήματα που ισχύουν σε ένα κράτος μέλος. Είναι σαφώς αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μόνο όταν αφορά θέματα οικογενειακού δικαίου που έχουν διασυνοριακό χαρακτήρα. Και είναι ένα από τα θέματα όπου θα ισχύει η ομοφωνία στο Συμβούλιο. Όσον αφορά το ερώτημα της κυρίας Σίγκβελτ, έχετε δίκιο για κατά το μεγαλύτερο μέρος δεν είναι νέοι τομεί ε, δραστηριότητα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι τομεί όπου η συνθήκη τη Λισαβόνα θα διευκρινίσει το βαθμό των αρμοδιοτήτων. Και δεν θα αφήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση να μπει σε νέους τομείς ενώ το άρθρο 308 τώρα επιτρέπει στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα να περάσει σε κάποιου τομεί πολιτική όταν δεν υπάρχει κάτι άλλο. Επομένω θα είναι διευκρίνηση και σε κάποιο βαθμό και περιορισμό του εύρου των δραστηριοτήτων ε, από τι δύο προηγούμενε συνθήκε. Όπω είπε ο συνάδελφο κύριο Σπερίλο, ευχαρίστω να επανέλθουμε και να απαντήσουμε στην Επιτροπή σας σε άλλες ερωτήσεις. Και όσον αφορά το χειρόφρονο που αναφέρατε από κάποιο κράτος μέλος που δεν θα δεσμεύεται από μια απόφαση, αν μπορεί δηλαδή ένα κράτο μέλο που δεν δεσμεύεται να μπλοκάρει μια απόφαση, και αυτό θα το εξηγήσουμε και αν η Επιτροπή, μας, ε, και αν η Επιτροπή το επιθυμεί να επανέλθουμε να δώσουμε την απάντησή μα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μπράντλεϊ. Κύριε Νίλσον από την Σουηδική Προεδρία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολύ σύντομα για τις τρεις ερωτήσεις που απευθύνθηκαν προς εμένα. Καταρχήν ε, για τα στοιχεία επιβατών, τα PNR στο Συμβούλιο αλλά και στο Κοινοβούλιο πιστεύω η κατάσταση είναι τέτοια που δεν σκεφτήκαμε να συνεχίσουμε τις συζητήσεις. Δεν θα συνεχίσουμε τις συζητήσεις στο Συμβούλιο. Θα περιμένουμε τη νέα συνθήκη της Λισαβόνας και όταν τεθεί σε ισχύ θα δούμε αν η Επιτροπή καταθέσει νέα πρόταση. Όμως για τα στοιχεία επιβατών θα ήθελα να τονίσω ότι ποτέ δεν ετέθη θέμα του αν θα πρέπει να χρησιμοποιούμε τα στοιχεία επιβατών ή όχι, διότι νομίζω ότι το PNR χρησιμοποιείται στα περισσότερα κράτη-μέλη. Όπω είπε ο υπουργό μου εδώ στο Κοινοβούλιο, περίπου 80% όλων των κατασχέσεων ναρκωτικών που γίνονται σε αεροδρόμια γίνονται χάρη στο σύστημα PNR. Η υπουργό μα ε, είναι πεπισμένοι για την χρησιμότητα του σύστηματο PNR. Όσον αφορά ε, το αν ήρθαμε σε επαφή μαζί σας κυρία Ιγκβελτ ε, για την έκθεση της Europol Ευχαριστώ να έρθουμε σε επαφή μαζί σας και να αρχίσουμε να σας καλέσω σε γεύμα και να αρχίσουμε να το συζητάμε να συζητάμε τα θέματα της Europol και σε οποιονδήποτε άλλο, ε, σε οποιοδήποτε άλλο μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αν δεν έχουμε έρθει ε, σε επαφή μαζί σας, σας διαβεβαιώνω ότι θα έρθουμε σε επαφή μαζί σας το συντομότερο δυνατόν, ούτως ώστε να κάνουμε τις σχετικές συζητήσεις. Σχετικά με το SWIFT, ήδη παρουσιάσαμε τη θέση μας για το SWIFT εδώ στο Κοινοβούλιο και δίπλα μου κάθεται και ο πρόεδρος της Επιτροπής ε, που ασχολείται με αυτό το θέμα και έχει έρθει δύο φορές στο Κοινοβούλιο. Εδώ έχουμε μια προσωρινή συμφωνία 12 μηνών και ίσως και λιγότερο. Και ο στόχος αυτής της συμφωνίας θα είναι να μην σταματήσουμε τις πολύ χρήσιμες πληροφορίες που λαμβάνουμε σύμφωνα με το αποκαλούμενο σύστημα TFTP για να μπορούμε να εμποδίζουμε τρομοκρατικές επιθέσεις και στην Ευρώπη. Πράγμα το οποίο έχει ήδη γίνει και είμαστε πεπισμένοι ότι η Επιτροπή θα δώσει νέα εντολή διαπραγματεύσεων ε, όταν θα τεθεί σε ισχύ η συνθήκη της Λισαβόνας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Δεν θέλω να ξανανοίξω τη συζήτηση αλλά έχω την εντύπωση ότι η κυρία Ινβέλτ θα ήθελε να ακούσει από την Προεδρία κάποιε διευκρινήσει. Μα, μα ήλπιζα ότι θα δεχόταν την πρόσκλησή μου για μεσημεριανό φαγητό. Είναι πάρα πολύ ρομαντικά όλα αυτά, λέει η κυρία Ινβέλτ. Ωραία, ωραία. Δεν δέχομαι. Δέχομαι. Ο, κοιτάξτε, όσον αφορά το PNR θα ε, έρθω σε επαφή μαζί σας σε διμερή βάση, κατηδίαν. Λοιπόν, δεν ε, θα προχωρήσουμε περισσότερο αυτή τη στιγμή και στρεφόμαστε πάλι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κυρία Κοράδο. Ίσως να ξεκαθαρίσω κάτι το οποίο αναφέρθηκε σε σχέση με αυτήν την ανακοίνωση Omnibus και τις εκρεμείς προτάσεις. Ε, ε, δεν θα καλυφθούν μόνο οι προτάσεις του πρώτου πυλώνα Πράγμα που σημαίνει ότι για τα μέσα τα οποία κρεμούν ενώπιον της Επιτροπής σας, εδώ είναι μόνο λίγα μέσα ε, για την ε, μετανάστευση, τις μακροχρόνιες θεωρήσεις ή κάποια θέματα Σέγγεν. Αλλά πάντως ε, δεν ε, δεν είναι πολλά, πολλοί φάκελοι. Οι περισσότεροι φάκελοι είναι ε, νομοθετικές προτάσεις τρίτου πυλώνα. Και άποψη επιτροπής είναι ότι αυτές οι εκκρεμείς προτάσεις, εάν δεν έχουν εγκριθεί ε, επίσημα και δεν έχουν δημοσιευθεί πριν από θέση ισχύ της νέας συνθήκης, τότε θα καταπέσουν, δεν θα υπάρχουν πλέον αν θέλετε, και θα πρέπει να υποβάλουμε νέες προτάσεις με βάση τη νέα νομική βάση. Θα το πράξουμε, αλλά επειδή τώρα έχουμε τη μετάβαση προς μια νέα επιτροπή και νέους επιτρόπους, οι πολιτικές αποφάσεις θα πρέπει να ληφθούν από τη νέα Επιτροπή. Και φυσικά η συζήτηση θα είναι ενδιαφέρουσα και ε, με το Κοινοβούλιο για τις προτεραιότητες. Και βεβαίως όλοι περιμένουμε με υπομονησία να δούμε τη συζήτηση αυτή. Finally, it might be to... Ευχαριστώ. Τέλος, ίσως ήταν χρήσιμο να ακούσουμε ε, την κυρία Ντανιέλ Ρεσάρντ για να μας ενημερώσει για τους πόρους που είναι διαθέσιμοι. Για τα τεχνικά σημεία, τα νομικά θέματα που, έχουν, που θίγουν διάφορα ερωτήματα τα οποία πρέπει να απαντηθούν. Έχετε το λόγο. Merci, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πράγματι, ε, τύχει ε, για την υπηρεσία μου να ε, βρίσκεται σήμερα εδώ που μιλάμε για την οδό που θα πρέπει να ακολουθήσουμε για την ενόψη της έγκρισης ε, της και της εφαρμογής συνθήκης Λισαβόνας. Αυτό σημαίνει ε, πολλά νέα θέματα ε, και έρευνα που απαιτείται και εμείς είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Στην προηγούμενη θητεία απαιτήθηκε πολύς χρόνος έτσι ώστε τα μέλη και οι επιτροπές να ενημερωθούν για τις υπηρεσίες που μπορούν να τους ε, ε, προσφέρουν τις μονάδες έρευνας, τα τμήματα έρευνας. Κοιτάξτε, κάθε κοινοβουλευτική επιτροπή έχει στη διάθεσή της ένα κάποιο προπολογισμό για έρευνα ανεξάρτητα από τις υπηρεσίες της γραμματείας για τη διαχείριση των εργασιών της Επιτροπής. Όσον αφορά την Επιτροπή σας, ε, το δικό μου τμήμα, η δική μου μονάδα, ε, θεματικό τμήμα ε, δικαιώματα των, ε, των πολιτών και συνταγματικά θέματα. Εμείς καλύπτουμε και τις αδελφές επιτροπές νομικών θεμάτων, αναφορών, γυναίκας και συνταγματικών υποθέσεων. Το θεματικό τμήμα, στη δική σας περίπτωση, ε, διαθέτει τρει εμπειρογνώμονε που κάθονται εδώ δίπλα μου, Αλεσάνδρο Νταβολή, Ζαν Λοή Αντουάν Γκρεγουάρ και Έλεν Κάλερς, που εργάζονται ο πρώτο σε θέματα προστασία δεδομένων αστυνομική συνεργασία και δικαστική συνεργασία σε ποινικέ υποθέσει. Ο δεύτερο συνάδελφο σε θέματα ε, ε, θεμελιώδη δικαιώματα και δικαίωμα ασύλου. Ε, και η συνάδελφο πολιτική ε, παράνομη και νόμιμη μετανάστευση, άσυλο, διέλευση εξωτερικών συνόρων. πραγματοποιούμε λοιπόν εργασία έρευνα είτε αναθέτω εξωτερικά ορισμένε έρευνε, κυρίω όταν είναι συγκρι... Ε, ε, συγκριτικέ και μακρόπνοε, που και δεν έχουμε εμεί τα μέσα, σε αυτή την περίπτωση συνεργαζόμαστε με ερευνητικά Ινστιτούτα σε όλη την Ευρώπη ε, μέσω προκήρυξης ε, ε, υποβολής προσφορών και υιοθετώντα την πρόταση μας φαίνεται ότι θα μας οδηγήσει στις απαντήσεις που θέλετε κι εσείς. Και πάντα στο μέτρο των πόρων μας και των υλικών και ανθρώπινων προσπαθούμε να αντιμετωπίζουμε και ορισμένες έρευνες σε εσωτερικό επίπεδο. Πρόκειται για επιστημονική εργασία με στόχο ε, την εξέταση σε βάθος που δεν μπορεί να αφορά απαραίτητα μία, διαδικαστική, μία διαδικασία κοινοβουλευτική, μπορεί να καλύπτει περισσότερες. Π.χ. αυτή τη στιγμή, από την προηγούμενη θητεία, έχουμε ζητήσει δύο μεγάλες μελέτες. Η πρώτη για την κατανομή του βάρου σε θέματα ασύλου και η άλλη για το κοινό καθεστώς ασύλου που θα αποτελέσει και προτεραιότητα της Επιτροπής σας ε, στην αρχή της νέας θητείας σας. Για να μπορέσετε να καταλάβετε τι κάνει η θεματική υπηρεσία μας και να καταλάβετε τι μέσα προσφέρουμε, έχουμε αυτά τα ογκώδη ντοσιέ, τα οποία έχετε μπροστά σας ε, και αυτή ε, η μέθοδος ε, κατά την άποψή μα, κοιτάξτε, ε, είναι, ε, την κάνουμε μόνο για τι δικέ μα τι επιτροπέ, είναι ασυνήθιστη αυτή η μέθοδο. Πάντω παρουσιάζει το εξή τριπλό πλεονέκτημα. Ότι είναι εξατομικευμένη, γιατί εμεί κατα... λάβαμε υπόψη το προσωπικό σα προφίλ, ε, γλωσσικέ σα ικανότητε κτλ. Όχι δηλαδή μόνο τη μητρική σα γλώσσα, αλλά και τη δεύτερη γλώσσα που γνωρίζετε, για τα έγγραφα τα οποία δεν υπάρχουν σε όλε τι γλώσσε εξατομικευμένο μέσο που μπορεί να εξατομικευτεί περαιτέρω. Δηλαδή ελπίζουμε ε, να αφαιρέσετε ότι δεν σας ενδιαφέρει και να συμπληρώσετε αυτά που σας ενδιαφέρουν. Και ε, πρόκειται για, ένα δυναμικό μέσο γιατί ε, όσο θα εγκρίνονται ορισμένα κείμενα, παράδειγμα νομοθεσία σε θέματα ασύλου, το Α ή το Β τμήμα του ντοσιέ θα αντικατασταθεί από το Α ή το Β νέο τμήμα ή θα προσθέσουμε ορισμένα στοιχεία τα οποία είναι σημαντικά. στην τελευταία ανάλυση εσείς είσαστε ε, αυτοί που θα αποφασίσετε για την τύχη του συγκεκριμένου ντοσιέ. Και θα δείτε πώς θα συλλέγετε εκεί τις βασικές πληροφορίες. Συμπληρώνεται και με κάποια πιο σύγχρονα εργαλεία, CD-ROM για τα τεχνικά δελτία και ένα κλειδί USB. Άρα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις μεθόδους. Η εμπειρία ε, έχει δείξει ότι ε, το USB το χρησιμοποιεί κανείς για να τυπώνει διαρκώς. Άρα καλό και το δοσιέ για να ε, αποθηκεύετε αυτά τα οποία θα τυπώνετε. Είναι, ε, είναι κάτι το οποίο το κάνουμε για πρώτη φορά και μόνο για ορισμένες κοινοβουλευτικές επιτροπές. Διευκρινίζω ότι αν δεν μπορείτε να πάρετε το ντοσιέ σας γιατί πρέπει να φύγετε, μπορείτε να το δώσετε στους κλητήρες που το πάνε στο γραφείο σας. Ε, περιμένουμε τα δικά σας σχόλια, το δικό σας feedback. Διευκρινίζω ταυτόχρονα ότι για λόγους ελέγχου ε, χρήσης των δημοσίων πόρων, όταν ένα μέλος ε, θέλει η μονάδα μας να ασχοληθεί με μία έρευνα, πρέπει να περάσει από τους συντονιστές που θα πάρουν απόφαση και που ενδεχομένως έχουν θέση και προτεραιότητες. Αυτό θέλω να πω και ευχαριστώ. Ευχαριστώ ε, για αυτά που μας είπατε κυρία Ρισάρ. Ερωτήσεις για αυτά τα θέματα. Ο κ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι απλό το ερώτημά μου. Βλέποντα αυτό που έχω μπροστά μου, ρωτώ το εξή. Ρωτώ την κυρία Ρισάρ. Εάν πράγματι στο θέμα, το θέμα της παράνομης μετανάστευσης. Θα τον... Της λαθρε... λαθρομετανάστευσης. Τι τίτλο θα δώσουμε, λαθρομετανάστευση ή παράνομη μετανάστευση. Γιατί και από νομική άποψη ε, η όρη είναι διαφορετική. Και εδώ εμείς που είμαστε στην προηγούμενη θητεία, τουλάχιστον εγώ, το φαινόμενο αυτό το ονομάζω παράτυπη ή λαθρέα μετανάστευση. Αλλά σε πολλά κείμενα εξακολουθώ να βλέπω τον όρο παράνομη μετανάστευση. Σας παρακαλώ να μου εξηγήσετε τι γίνεται. Γιατί θα πρέπει όλοι να μιλάμε για το ίδιο πράγμα. Τουλάχιστον σε τέτοια στοιχειώδη ζητήματα να ακολουθούμε του ίδιου όρου. Κύριε Ρησάρ, για το θέμα αυτό. στο μέτρο που υπάρχει συνένεση, ε, συμφωνούμε απόλυτα. Να αλλάξουμε τον όρο. Δεν ξέρω σε ποια γλώσσα. Σε, τι έχετε, ποιο είναι το πρωτότυπο που έχετε. Στα αγγλικά είναι irregular immigration. Και legal migration που αντιστοιχούν βέβαια σε διαφορετικές βάσεις της συνθήκης και στα γαλλικά και σαφώ ε, υπάρχει μια διαφορά. Εάν έχετε μια σαφή άποψη συνενετική μπορούμε να αλλάξουμε τον όρο. Να, μα γι' αυτό σας λέω ότι πρέπει να ενημερώνουμε διαρκώς το ντοσιέ. Κύριε Ρισάρ, δεν ξέρω κατά πόσο υπάρχει συνένεση και τι γίνεται με τη συνθήκη της Λισαβόνας. Δεν ξέρω τι σχέση έχει. Δεν ξέρω τι επίσης ορολογία ακολουθούμε στην συνθήκη της Λισαβόνας. Γιατί η βάση της νομικής συνένεσης θα είναι η συνθήκη της Λισαβόνας. Κύριε Δίας Δεμέρα. Θέλετε να πείτε κάτι. Ναι κύριε Πρόεδρε. Ένα μικρό σχόλιο για να ξεκαθαρίσω κάπως. Γιατί έχω αμφιβολίες. Θέλω να πω ότι εδώ δεν βρισκόμαστε απέναντι μόνο σε μια νομική έννοια, αλλά και σε, μια πολιτική, σε ένα πολιτικό όρο. Είναι σύνηθες σε όλες τις εκθέσεις μας, στην προηγούμενη θητεία, όταν μιλούσαμε για μετανάστευση, συγκεκριμένες πολιτικές ομάδες μιλούσαν για παράνομη μετανάστευση, ενώ άλλες πολιτικές ομάδες μιλούσαν για παράτυπη μετανάστευση ή για ε, λάθρο μετανάστευση. Πέραν τούτου, μάλλον ξέρετε από αυτό, και να σα πω το εξή, θα μιλήσω για μια οδηγία που είναι πολύ προβληματική για ορισμένου, ενώ για άλλους είναι πολύ απαραίτητη. Την οδηγία για την επιστροφή. Εκεί αναφέρεται σαφώ ο όρο παράνομη μετανάστευση. Παρανομή. Και εγώ σα λέω τώρα ποια είναι η θέση μου. Η θέση μου είναι ότι θα πρέπει να την ονομάζουμε παράτυπη ή λάθρο μετανάστευση. Και ανεξάρτητα με τι απόψει των μεν και των δε διάφορε ομάδε. Δεν είναι νομική μόνο η έννοια, είναι και ιδεολογική φύσεω η διαμάχη. Και όσον αφορά την κυρία Ρισάρ, τη λέω το εξή. Το αντίθετο τη παράτυπη ή λαθρέα μετανάστευση δεν είναι η νόμιμη, γιατί όπως σας είπα και το ξαναλέω, εδώ μιλάμε και ιδεολογικέ φύσης διαφορές και όχι μόνο νομικέ. Για να δούμε μήπως μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ε, ένα κοινό όρο και να συνεννοηθούμε. Ευχαριστώ. Πριν δώσω, πριν πάμε στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης, φαίνεται το κύριο Μπουσούτιλ. Κύριε Μπουσούτιλ, να προσθέσετε κάτι. Όχι, θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω τους ε, εκπροσώπου τη Νομική υπηρεσία για την παρουσίασή τους και έχω να ρωτήσω ε, το εξή. Σωστά αντιλαμβάνομαι ότι πέρα από την δουλειά τους υπάρχει και ένα επιπρόσθετος προπολογισμό για την Επιτροπή μα, ώστε να μπορεί να κάνει μελέτες ανεξάρτητα από ε, το τμήμα. Ε, ε, σωστά το αντιλαμβάνομαι αυτό. Και τι προϋπολογισμό έχουμε, θα μπορούσαν να μας πούν. Ένα δεύτερο ερώτημα. Τι μελέτες κάθε χρόνο μπορεί να παρέχει αυτό το τμήμα. Υπάρχει κάποιο όριο ετησίως, γιατί φαντάζομαι ότι δεν μπορούν να εκπληρώσουν όλες τις επιθυμίες για κατάρτιση μελετών. Και τέλος, πάντοτε περιμένουν οδηγίες από κάποια επιτροπή για να μπορούν να ξεκινήσουν μια έκθεση ή κάνουν και, θα λέγαμε, ιδία πρωτοβουλίας εκθέσεις. Ευχαριστώ. Κυρία Χισάχ, μπορείτε να διευκρινίσετε τις ερωτήσεις του κυρίου Μπουζουτήλ. Μάλιστα. Ναι, τρία σημεία. Λοιπόν, ναι, η Επιτροπή Ελευθεριών έχει προπολογισμό, όπως και οι άλλες επιτροπές. Μάλιστα αυξήθηκε πολύ ο προπολογισμό αυτός, που δεν είναι βέβαια εξαιρετικός, εάν λάβουμε υπόψη μας το προπολογισμό μελετών της Επιτροπής, αλλά που όμως μας επέτρεψε τα τελευταία χρόνια να ε, κάνουμε σημαντικές μελέτες. Ε, τώρα, το εάν υπάρχουν θεματικές ενότητες, τι να σας πω, ε, δεν μπορώ να απαντήσω 100%. Ε, δηλαδή, κύριε Βουζουτήλ, τι εννοείται, πέρα από τις εσωτερικές μας, από τους εσωτερικούς μας πόρους, εάν έχουμε δυνατότητα να κάνουμε και την αρμοδιότητα και τα χρήματα να κάνουμε κάποιες μελέτες, τις κάνουμε. Απ' την άλλη πλευρά όμως ζητούμε και από εξωτερικούς φορείς να διεξάγουν Μελέτε μελέτες ε, για ε, λογαριασμό μας. Τρίτον, ε, δεν ξεκινούμε με δικιά μας πρωτοβουλία, αλλά πάντοτε μετά από αίτημα των ε, ε, κοινοβουλευτικών επιτροπών και για τις μελέτες που κάνουμε εμείς οι ίδιοι, αλλά κυρίως όταν πρόκειται για δαπάνη δημοσίου χρήματος. Δηλαδή μπορούμε να δεσμεύσουμε χρήματα μονάχα και εφόσον υπάρχει συγκεκριμένη απόφαση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών Ας πούμε, εάν κάποιος βουλευτής θέλει να ασχοληθούμε με κάποιο συγκεκριμένο ζήτημα, θα πρέπει να προωθήσει το θέμα στην Επιτροπή, ε, στη συνεδρίαση των συντονιστών και μετά από αίτημα αυτής ε, της ε, Επιτροπής των Συντονιστών μπορούμε εμείς να χρησιμοποιήσουμε οικονομικούς ή φυσικούς πόρους. Απήντησα ή ανθρώπινους πόρους. Ναι, Μπουζούτιλ, εγώ ήθελα να ξέρω εάν υπάρχει ανεξάρτητος προϋπολογισμός για την Επιτροπή μας ε, πέρα από, τους, από τον συνολικό προϋπολογισμό και από ό,τι κατάλαβα η απάντηση είναι όχι. Ε, πρόκειται για ένα συνολικό προϋπολογισμό για τις Επιτροπές. Αυτά. Σας ευχαριστούμε κύριε Ρουσά. Τώρα είναι ώρα να περάσουμε στα σημεία 5 και 6, τα οποία είπαμε ότι έχουν συγχωνευθεί. Πρόκειται ε, για κοινή συζήτηση για τη θέσπιση μηχανισμού αξιολόγηση για την επαλήθευση τη εφαρμογή του κεκτημένου του Σέγγεν, καθώ επίση και για το μηχανισμό αξιολόγηση για την επαλήθευση της εφαρμογής του κεκτημένου Σέγγεν. Θα ξεκινήσουμε με τον εισηγητή, τον κύριο Κάρλο Κοέγιο και μετά θα δώσουμε το λόγο στην Επιτροπή και ε, στο Συμβούλιο, ε, στους αντιπροσώπους τους δηλαδή. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Για κύριο Σκοαγιο. Πρώτα απ' όλα πρέπει να πω ότι είμαι πολύ ικανοποιημένος ε, για την πρωτοβουλία αυτή που ε, θέλει να κάνει τον μηχανισμό αξιολόγησης ε, της εφαρμογής του κεκτημένου Σέγγεν πιο συνεκτικό αλλά και πιο απλό και πιο διαφανή μηχανισμό. Ε, δυστυχώς δεν διαφαίνεται αυτό από τις προτάσεις που μας υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όντως, ε, οι, επιτροπή, οι προτάσεις αυτές ε, έχουν έναν και μόνο νεοτερισμό. Ε, δηλαδή ότι μπορούμε να προχωρήσουμε σε μη σε επισκέψεις, πράγμα το οποίο θεωρούμε απολύτως θετικό. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει στόχο την μεταβίβαση ε, της, ε, των όσων έκαναν μέχρι τώρα τα κράτη-μέλη ε, σε αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και βεβαίως πρέπει να πω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ήταν μάλλον ξένο προς την διαδικασία αξιολόγησης του κεκτημένου Σέγγεν. Πρέπει να πω ότι δεν συμφωνώ με τον τρόπο προσέγγισης. Πρώτον, υπάρχει διαχωρισμός της εντολής, δηλαδή αξιολόγηση των χωρών πριν την είσοδό τους στο Σέγγεν ε, και τις χώρες που βρίσκονται ήδη ε, στον χώρο Σέγγεν. Πρόκειται για μία ε, κίνηση η οποία σημαίνει οικονομικό βάρος. Δεν χρειάζεται αυτός ο διαχωρισμός. Δεύτερον, όσον αφορά την μεταβίβαση των δεδομένων. Δεν χρειάζεται να μπω σε υπερβολικές λεπτομέρειες, αλλά πρέπει να σας πω ότι ας πούμε δεν γίνεται λόγος για το outsourcing, την προσφυγή δηλαδή στις υπηρεσίες εξωτερικών παραγόντων. Ε, επίσης, ε, δεν γίνεται λόγος για το σύστημα VIS και επίσης για τους ε, οικονομικούς ελέγχους και για τις ε, ε, εκθέσεις επιθεώρησης δεν γίνεται σωστή αξιολόγηση. Πέρα όμως από αυτά τα τυπικά υπάρχει και ένα θέμα ουσίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε μελετήσει το θέμα αυτό στις προηγούμενες θητείες ε, προσφεύγοντας στην ε, γνώμη της νομικής υπηρεσίας, δηλαδή ε, να μελετήσει το κατά πόσον η νομική βάση ήταν σωστή ή όχι. Η απάντηση λοιπόν της νομικής υπηρεσίας είναι εξή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να παρουσιάσει, να υποβάλει πρωτοβουλία βάσει αυτής της νομικής βάσης που θα ζητάει μονάχα την διαβούλευση του Κοινοβουλίου, αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τροποποιώντας το βασικό κανονισμό που έχει ήδη εγκριθεί σε διαδικασία συναπόφαση με το Κοινοβούλιο. Θα μπορούσε λοιπόν, λέγω, η Επιτροπή να περάσει σε συναπόφαση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εάν και οι δύο ε, λύσεις ήταν ικανοποιητικές γιατί επέλεξε μία από τις δύο η Κομισιόν για λόγους πολιτικούς γιατί θεώρησε ότι δεν θα έπρεπε να δώσει στο Κοινοβούλιο την δυνατότητα της συναπόφασης. Όσον αφορά τώρα ε, την εφαρμογή του συστήματος ε, Σέγγεν νομίζω ότι πολλά μπορούμε να πούμε όσον αφορά το σύστημα αμοιβαίας εμπιστοσύνης από τη στιγμή που δεν υπάρχουν έλεγχοι στα σύνορα μπορούμε να φανταστούμε ότι οι, ε, ότι έλεγχοι θα γίνονται στα εξωτερικά σύνορα από μια δεδομένη χώρα ε, και επομένως οι έλεγχοι αυτοί θα πρέπει να θεωρούνται ικανοποιητικοί. Εδώ κράτησε κάποιες επιφυλάξει η Επιτροπή και οι χώρε μέλη επίσης. Και εδώ βεβαίω και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μια και εκπροσωπεί του Ευρωπαίου ψηφοφόρου θα πρέπει να έχει το λόγο του όσον αφορά το θέμα αυτό, γιατί πρόκειται για ζητήματα τα οποία αφορούν άμεσα ε, τους ε, πολίτες ε, της Ευρώπης μιλάμε για συγκεκριμένες αρμοδιότητες ε, οι οποίες θα πρέπει να εφαρμόζονται με τρόπο ε, σωστό κυρίως όταν, αφορά, ε, όταν αφορούν βασικά νομικά κείμενα. Πρέπει να υπενθυμίσουμε κύριε Πρόεδρε επίσης και εφόσον εφαρμοστεί η συνθήκη της Λισαβόνας όλα αυτά τα εργαλεία θα πρέπει να ευθυγραμμιστούν με τη νέα συνθήκη και άρα τι θα πρέπει να κάνουμε θα πρέπει να προβλέψουμε την απόρριψη αυτών των πρωτοβουλειών Λοιπόν, θα πρέπει να καλέσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποσύρει τις πρωτοβουλίες αυτές και να υποβάλει καινούριε. Και σύμφωνα με αυτά που λέει και η έκθεση, να τα υποβάλει τα νέα αιτήματα και τις νέες πρωτοβουλίες σύμφωνα με τη διαδικασία της συναπόφασης. Και με τον τρόπο αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα παίξει πολύ, πολύ σημαντικότερο ε, ρόλο στα νέα, στους νέους αυτούς μηχανισμούς για την αξιολόγηση Σέγγεν. Αυτά. Θέλει ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, να πάρει το λόγο. Είναι η εκπρόσωπος. Uh, Σας ευχαριστώ. Όσον αφορά, όσον αφορά τα σημεία αυτά, νομίζω ότι η πρόταση της Επιτροπής δεν είναι η απλή εισαγωγή αυτών των μη αναγγελθέντων ε, επισκέψεων, αλλά αναφέρει και άλλους μηχανισμούς στη φάση της παρουσίασης ε, ε, του διορισμού εμπειρογνωμόνων που συμμετέχουν στους αξιολόγηση κλπ. Επίσης, η Επιτροπή έχει την άποψη ότι δεν υπάρχει επικάλυψη ανάμεσα στο πρώτο τμήμα της τρέχουσας εντολής και στο δεύτερο, διότι σε κάποιο στάδιο οι αξιολογήσει πριν από, πριν από την άρση ε, των εσωτερικών ελέγχων θα ε, τείνουν να μειώνονται γιατί αυτή τη στιγμή τρία κράτη-μέλη δεν είναι μέλος ε, της, ε, του, του, του Σέγγεν χωρίς, με, με, άρση, με εξάλληψη δηλαδή των εσωτερικών ελέγχων. Όπω είπε τώρα και ο εισηγητή, έχουμε τι εξή πιθανότητε ω αφορά την νομική βάση. Το άρθρο 66 και ε, να στηρίξουμε από την άλλη αυτή την πρόταση ε, στις ουσιαστικές, στις ουσιαστικές νομικές βάσεις. Εμείς καταλήγουμε σε πέρασμα ότι το 66 είναι ε, η σωστή βάση. Διότι ο μηχανισμός αξιολόγησης του Σέγγεν δεν αλλάζει το ουσιαστικό και εκτιμένο. Με αυτές τις προτάσεις δεν τροποποιούνται, για παράδειγμα, οι συνθήκες εισόδου, ε, δεν αλλάζουν οι προϋποθέσεις ε, για χορήγηση ή θεώρησης. Γι' αυτό Επιτροπή στήριξε την πρότασή της στο άρθρο 66. Παρ' όλα αυτά, η Επιτροπή συνειδητοποιεί ότι πρέπει να συμμετέχει πιο στενά ε, το Κοινοβούλιο σε αυτό το μηχανισμό και αυτό αντικατοπτρίζεται και στην πρόταση, όπως για παράδειγμα η υποχρέωση υποβολής έκθεσης στο Κοινοβούλιο. Όσον αφορά το μέλλον, όταν δηλαδή θα αρχίσει να ισχύει η συνθήκη της Λισαβόνας, όσο δεν έχει ε, τεθεί σε ισχύ, ε, ε, θα, πρέπει να εργαστούμε με την υφιστάμενη νομική βάση. Στη συνέχεια όμως και αυτές οι προτάσεις θα συμπεριληφθούν στη δήλωση Omnibus όπως ήδη αναφέρθηκε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Λέγομαι Χρήστο Χέμπορντ και είμαι προεδρεύων της ε, ομάδος αξιολόγησης του Σέγγενε υπό την Σουηδική Προεδρία. Ξεκινήσαμε λοιπόν την αναθεώρηση του κανονισμού ε, που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα συνεχίσουμε αύριο, ε, γιατί είχαμε σταματήσει τα άρθρα 9 και αύριο θα συνεχίσουμε τα άρθρα 10 έως 18 πέρα από το τι θα συμβεί τελικά ή στο μέλλον, εμείς πιστεύουμε ότι είναι χρήσιμο να αποσαφηνίσουμε τη θέση των κρατών ε, μελών όσον αφορά συγκεκριμένα, ε, τα συγκεκριμένα άρθρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σα the members, Σας ευχαριστώ πολύ. Τα μέλη τώρα, κύριος De Jong. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Βεβαίως μπορώ να συγχαρώ τον ε, εισηγητή για την προσέγγιση την οποία ακολούθησε και που βρίσκει απολύτω σύμφωνη την πολιτική μας ομάδα. Και πραγματικά στηρίζομαι και την ε, ε, πρότασή του να δεχτεί την νομική αυτή βάση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κάτι άλλο. Κοιτάζοντας προσεκτικά και επί της ουσίας την έκθεση υπάρχει ένα θέμα το οποίο δεν αναφέρεται στο παράρτημα ε, που, ε, όπου καταγράφονται όλα τα σημεία τα οποία θα πρέπει να συζητηθούν και να επαληθευθούν. Η ομάδα μας έχει ένα πρόβλημα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο γίνεται λόγος για τον έλεγχο των συνόρων, κυρίως όσον αφορά τα θέματα που άπτονται των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν ξέρω πώς εφαρμόζεται το δικαιοκτημένο του Σέγγεν, αλλά όπω και αν εφαρμόζεται, δεν είναι δυνατόν να αγνοήσει κανεί ότι ό,τι και αν κάνει και με όποιο τρόπο και αν το κάνει πρέπει να σέβεται τα, τα ανθρώπινα ε, δικαιώματα και επομένω θα πρέπει να υπάρξει ξεχωριστό κεφάλαιο για το θέμα αυτό στο παράρτημα. Να πω τέλος ότι πρόκειται για μια ουσιώδη συζήτηση και ε, ότι οπωσδήποτε στηρίζομαι πλήρως τον εισηγητή. Ε, και θέλουμε λοιπόν να γίνει επαναυποβολή του θέματος με τη σωστή νομική βάση. Ευχαριστώ. Η κυρία Λάτφορντ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Κοέγιο για την ε, σωστή έκθεση του η οποία βασίστηκε σε συζήτηση, ε, σε βάθος ανταλλαγή απόψεων και στην Επιτροπή μας για θέματα Σέγγεν κλπ. έθιξε ορισμένα ε, ζητήματα ε, στην πολύ ενδιαφέρουσα και χρήσιμη έκθεσή του που αντικατοπτρίζουν ακριβώς τις συζητήσεις που κάναμε και εδώ. Ε, είμαι ευγνώμων στον κύριο Κοέγιο γιατί απομόνωσε και κάποια σημεία τα οποία αφορούν την εφαρμογή του συστήματος πληροφοριών και που σχετίζονται και με αυτά τα οποία τελικά κατέληξαν στον ε, κωδικό θεωρήσεων, Visa Code, στον κώδικα συγγνώμη των θεωρήσεων, ε, Visa Code. και ε, ε, θυμάμαι μάλιστα ότι και σε ε, θέματα τα οποία σχετίζονται με, ασφάλεια, με την ασφάλεια και την παροχή βίζας και τα λοιπά, ο κύριος Κοέγιο είχε συζητήσει εντόνως και η συζήτηση που έκανε αντικατοπτρίζεται και στις προτάσεις που μας υπέβαλε. Άρα η έκθεση μας βρίσκει σύμφωνο, βρίσκει σύμφωνη την ομάδα μας και θεωρούμε θεωρούμε ότι η προσέγγιση του κυρίου Κοέγιο είναι σωστή και αξίζει τον κόπο να την ε, συζητήσουμε ε, με τη διαδικασία συν απόφασης. Ευχαριστώ. Μουράης. Um, Σα ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο σκιώδη μα δεν μπόρεσε να είναι παρόν. Απλά και μόνο θα ήθελα να μεταφέρω εκ μέρου του αυτά τα οποία είπε και η κυρία Λάτφουρ. Είμαστε ε, σε καλά χέρια με τον κύριο Κοέλιο σε αυτή την έκθεση και συμφωνούμε απόλυτα με την άποψή του όσον αφορά τη διαδικασία που ακολουθείτε. Πρέπει να έχουμε συναπόφαση. Και απλά και μόνο θέλω να καταγράψετε την άποψη τη ομάδα μου όσον αφορά το σημείο αυτό. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ. Να ξαναδώσουμε το λόγο στον κύριο Κοέλιο. Δεν έχω τίποτα άλλο να προσθέσω, Πρόεδρε. Νομίζω ότι μπορούμε να ψηφίσουμε αύριο. Πολύ ωραία. Συμφωνήσαμε και σημείο αυτό. Αύριο λοιπόν θα ψηφίσουμε στην έκθεση. Με ενημερώνουν ότι το επόμενο σημείο το σημείο 4 είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Γιατί όλοι θα θυμόμαστε ότι ήταν ο κύριος Ζήλιντο Κερκόφ ήρθε για πρώτη φορά στην Επιτροπή μας μόλις αναλάβουμε τη θητεία μας, είχαμε μια ουσιαστική ανταλλαγή απόψεων Αλλά δεν είχαμε χρόνο να προχωρήσουμε στη συζήτηση. Αναφέρθηκαν πολλά σημεία, αλλά δεν μπορέσαμε για λόγους ε, χρονικού περιορισμού να αναπτύξουμε τη συζήτηση περαιτέρω. Θα έρθει λοιπόν ακριβώς στις 5. Στις 5. Έχει προγραμματιστεί να έρθει. Επειδή λοιπόν αυτό θα είναι το επόμενο θέμα μας, Ίσως θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα και να επαναλάβουμε τις εργασίες μας σε 20 λεπτά ακριβώς, στις 5 η ώρα. Διάλειμμα λοιπόν τώρα.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 ver, maestro.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 Please, dear colleagues, take your seats. Καθίστε αγαπητοί συνάδελφοι για να ξαναρχίσουμε τη συνεδρίασή μας. Euh, Καλώς ήρθατε κύριε Ζιλ Ντεκέρχοφ. Ο κύριος Ζιλ Ντεκέρχοφ είναι ο συντονιστής της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με, τις, ε, με το πρόγραμμα δράσης για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Κάναμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση στην τελευταία παρουσίαση που μας είχε κάνει στην Επιτροπή μας στις 3 Σεπτεμβρίου. Δεν είχαμε το χρόνο για να κάνουμε όλη τη συζήτηση που θέλαμε και νομίζω ότι αξίζει τώρα να κάνουμε αυτή τη συζήτηση για τα θέματα του κ. Ντεκέρχοφ και του δίνω το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω θα ήταν προτιμότερο να κάνουμε μια ανταλλαγή απόψεων. Την προηγούμενη φορά εγώ προσπάθησα να εξηγήσω τους βασικούς άξονες της έκθεσής μου και τα στοιχεία της απειλής που μπορεί να υπάρχει και καλύτερα θα ήταν να ζητήσω από τους κυρίους και κυρίες βουλευτές να κάνουν ερωτήσεις και εγώ θα απαντήσω. Βεβαίω. Να ξεκινήσουμε λοιπόν, ο κύριος Χάρκε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Άκουσα αυτά που είπε ο κύριος Κέρχοφ στις αρχές Σεπτεμβρίου με μεγάλο ενδιαφέρον. Και θα ήθελα να πω ότι εκτιμούμε ιδιαίτερα τη δουλειά του, που είναι εξαιρετική, πολύ ποιοτική. Και νομίζω ότι χρειαζόμαστε μια επικαιροποιημένη νομοδότηση για την κατάσταση στα κράτη-μέλη στο πλαίσιο της αστυνομικής συνεργασίας και των πληροφοριών για το συντονισμό της αντιτρομοκρατικής δράσης. Μας είναι χρήσιμο να γνωρίζουμε το αν υπάρχει ομαλή ροή και αν η δική σας δουλειά μπορεί να συμπληρώνεται από τη δουλειά που γίνεται στα κράτη-μέλη. Θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι έστειλα μια επιστολή με βάση την παρέμβασή σας στις 3 Σεπτεμβρίου υπομορφή υποβολής παραπώνου και ζητώ την κατανόησή σας ε, για να κάνω και προφορικά την παρουσίαση αυτή. Τη συντάξαμε στις 9 Σεπτεμβρίου αυτή την επιστολή και μου κάνει εντύπωση γιατί δεν ξέρω πώς ε, η Επιτροπή... Εκεί λοιπόν συμπεριλαμβάνεται συνήθως η έκφραση ε, βασική ε, οργάνωση αποσχιστική για να παραπέμψει στην ε, τρομοκρατική έτα. Τότε είχα αναφέρει ότι θα μπορούσαμε να σκεφτούμε ότι ένα αυτόνομο όργανο της Επιτροπής θα μπορούσε να διαπράξει ένα τόσο σοβαρό σφάλμα, διότι Όσον αφορά το, ε, την, την, τον αγώνα κατά της τρομοκρατίας, ε, υπάρχει πρόβλημα με τους όρους και είναι πολύ ε, σοβαρό το να δημιουργείται σύγχυση όσον αφορά τους όρους αποτελεί βασικό στοιχείο της στρατηγικής του οργανισμού στον οποίο εσείς είστε επικεφαλής. Και θα ήθελα να υπενθυμίσω σε όλους ότι το να μιλάμε για την ΕΤΑ και να τις αποδίδουμε ε, τον πολιτικό όρο ότι πρόκειται για μια ε, οργάνωση ε, που αγωνίζεται για την απόσχηση είναι σοβαρό. Πολλοί υπερασπίζονται την ανεξαρτησία της χώρας των Βάσκων αλλά δεν δολοφονούν. Γι' αυτό το να χρησιμοποιούμε λοιπόν ένα πολιτικό όρο για τους δολοφόνους τότε καταλαβαίνετε ότι αξιολογούμε θετικά αυτή την τρομοκρατική οργάνωση και κάτι τέτοιο δεν μπορεί να το επιτρέπουμε. Είναι σαν την Αλκάιδα να την ονομάζαμε οργάνωση για την επέκταση του Ισλάμ. Η διάδοση του Ισλάμ. Το ήταν εξίσου σοβαρό. Πώ αισθάνονταν τα θύματα τη Αλκάιδα, ή πώ αισθανόμασταν πολλοί από εμά, ε, δημοκρατικοί πολίτε ε, τη χώρα των Βάσκων και τη Ισπανία, όταν βλέπουμε ότι ένα επίσημο όργανο κάθε ημέρα ε, στην, ε, ε, όταν αναφέρεται στην ΕΤΑ ως αυτονομιστική, ως αποσχιστική οργάνωση των Βάσκων. Θέλω λοιπόν δημόσια να εκφράσω την διαμαρτυρία μου. Gracias. Σας ευχαριστώ. Να μαζέψουμε κάπως ερωτήσεις. Και μετά μου κάνετε ερωτήσεις. Ο κύριος Μωράς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Δεκέρχοφ, ελπίζω να έχετε το χρόνο να απαντήσετε σε κάποιες από τις ερωτήσεις Τις θέτω και ελπίζω να βρείτε το χρόνο να απαντήσετε. Στο τέλος της προηγούμενης παρουσίασής σας, που ήταν πάρα πολύ χρήσιμη, δεν είχατε το χρόνο να μιλήσετε για την εθνοτική και θρησκευτική σύνθεση αυτών των ατόμων ε, και έγινε μια πολύ καλή ανάλυση για την, τον εθνοτικό ε, ε, χαρακτήρα και θα ήθελα να μας πείτε κατά πόσο αυτά τα στοιχεία λαμβάνονται υπόψη στις Έρευνε που γίνονται σε αεροδρόμια, παραδείγματο χάρη, είναι πολύ δύσκολο να γίνονται στατιστικές αναλύσεις και ε, θα ήθελα, ακόμη και αν δεν έχετε το χρόνο σήμερα να απαντήσετε, θα ήθελα να μου πείτε ότι είναι ένα θέμα που σας απασχολεί και το εξετάζετε, γιατί θέλουμε αποτελεσματικές λύσεις κατά της τρομοκρατίας. Δεν θέλουμε να δαπανούμε χρόνο και πόρου για να πιάνουμε λάθο. Ε, άτομα γιατί πολλές φορές μπορεί οι πληροφορίες για ε, το άτομο που ερευνάται να μην είναι ε, αυτές που οδηγούν στο στόχο μας. Μια δεύτερη ερώτηση τώρα για την πολιτική κατά της διαμόρφωσης ακραίων τάσεων. Ξέρω ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο, στη χώρα μου, έχουν γίνει σημαντικές πρόοδοι για το θέμα αυτό, για την καταπολέμηση των ακραίων τάσεων αλλά θα ήθελα να μας πείτε αν υπάρχει κάποια ισορροπία στα κράτη-μέλη για το πώς αντιμετωπίζουν αυτό το θέμα της ανάπτυξης ακραίων τάσεων. Νομίζω ότι δεν ε, είναι όλα τα κράτη-μέλη στο ίδιο επίπεδο όσον αφορά την διαμόρφωση πολιτικών κατά της, ε, κατά της ε, ανάπτυξης των ακραίων τάσεων. Ευχαριστώ πολύ κυρία Ευχαριστώ κύριε ε, Ντεκέρχοφ. Χαίρομαι ιδιαίτερα που ήρθατε στην Επιτροπή μας και έχω τρία συγκεκριμένα ερωτήματα. Πρώτον, νομίζω την περασμένη εβδομάδα το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για άλλη μια φορά ε, εξέδωσε μια απόφαση για το θέμα των blacklist και αποφάσισε ότι κάποιο μαχητή ε, υπέρ τη ελευθερία από τι Φιλιππίνε ή δεν ξέρω, μαχητή τη ελευθερία ή πώ αλλιώ θα τον ονόμαζε κανεί, έπρεπε να βγει από αυτόν τον κατάλογο, από αυτό, τον, ε, αυτό το blacklist. Και δεν είναι πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο. Ξέρω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάνει κάποιε ίσονο σημασία αλλαγέ στη διαδικασία θα έπρεπε να έχουμε διαδικασίες ε, που να αντιστοιχούν ε, σε μια δημοκρατία όπου κυριαρχεί το κράτος δικαίου. Μια δεύτερη ερώτηση. Επανειλημμένα ζητήσαμε μια εμπεριστατωμένη αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των πολιτικών για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Πότε θα μπορούσαμε να αναμένουμε αποτελέσματα μιας τέτοιας αξιολόγησης. Και τρίτη και τελευταία μου ερώτηση που είναι ευρύτερη για το πού εστιάζονται οι προσπάθειες καταπολέμησης της τρομοκρατίας. Διότι κάθε χρόνο οι εκθέσεις για την τρομοκρατία της Europol, παραδείγματος χάρη, δείχνουν ότι η πλειοψηφία των περιπτώσεων, πάνω από 95%, δεν είναι τρομοκρατία διακρατικού χαρακτήρα. Πρόκειται για αποσχιστικές ομάδες. Ε, φοβάμαι να μιλήσω με όρους, να μην ακουστεί λάθος όρος όταν λέω αποσχιστική. Τέλος πάντων, ε, κινήσεις ε, που είναι ενδεχομένως ακροδεξιές οργανώσεις ή νεοναζί, οργανώσεις νεοναζί και κάθε φορά που μιλάμε για τις πολιτικές καταπολέμησης της τρομοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνήθως επικεντρώνονται στην καταπολέμηση των ε, Ισλαμιστών ε, εξτρεμιστών. Δεν λέω ότι πρέπει να αποκλείονται, δεν ξέρω αν αυτή είναι η καλύτερη δυνατή κατανομή πόρων. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Ντεσαρίλ. <laughs> Ναι, σα ευχαριστώ. Καλησπέρα σα, κυρία Ντεκέρκοφ. Θέλω να σα ευχαριστήσω γιατί ήρθατε εδώ σήμερα και θέλω να σα πω ότι διάβασα με μεγάλη προσοχή τι εκθέσει σα για τη στρατηγική για την καταπολέμηση τη τρομοκρατία και για το πρόγραμμα δράση ε, ε, για την καταπολέμηση του φαινομένου αυτού. Και ευχαριστώ και τη Σουηδική Προεδρία που συμπεριέλαβε την Ευρωπαϊκή Συνεργασία ε, Καταπολέμηση Τρομοκρατία ε, ω προτεραιότητα. Τρει ερωτήσει θα ήθελα να σα κάνω σε σχέση με του πυλώνε στου οποίου στηρίζεται το πρόγραμμα δράση. Πρόληψη, δίωξη και απάντηση σε τρομοκρατικές πράξεις. Πρώτον, ε, σας προωθώ να ακολουθήσετε αυτόν τον κατάλογο στο πρόγραμμα δράσης, να καταπολεμήσετε την τρομοκρατία μέσω της έγκρισης μέτρων αποτροπής που παρεμποδίζουν ε, την, ε, τη δράση των εξτρεμιστικών ομάδων και την, ή άλλων ομάδων που στη συνέχεια μετατρέπονται σε τρομοκρατικές ομάδες. Εδώ τονίζω και το θέμα της εκπαίδευσης στο σχολείο και στην οικογένεια ως αποτελεσματικό μέσο για την αποφυγή κάθε μορφής ε, τρομοκρατίας, όχι μόνο διεθνούς αλλά και εθνικής. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω συγκεκριμένα, δεν πιστεύετε ότι θα χρειαζόμασταν ένα σαφή ορισμό της τρομοκρατίας. Γιατί χωρίς αυτόν τον ορισμό δεν μπορούμε να καταπολεμήσουμε το φαινόμενο αυτό, ούτε να το προλάβουμε ε, και στο διαδίκτυο και και στον τύπο ή και σε άλλο μέσο. Όσον αφορά τη δίωξη, εκφράζουμε την ικανοποίησή μα γιατί αυτή τη στιγμή ε, ε, ε πραγματικά υφίσταται πραγματική δίωξη οι τρομοκράτε. Αλλά υπάρχουν πολλοί τρομοκράτες που δεν εκδίδονται ε, και εξακολουθούν να διαπράττουν αδικήματα. Πώ μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτού του τρομοκράτε και πώ μπορούμε να του φέρουμε ενώπιον τη δικαιοσύνη. Γιατί επειδή εξακολουθούν να ζουν σε άλλε χώρε, ενώ είναι τρομοκράτε, ε, και υποστηρίζουν την τρομοκρατία. Αυτό αποτελεί σοβαρή ταπείνωση και απέναντι ε, στα θύματα. Και κάτι άλλο, θα μιλάτε για την απάντηση. Ξέρετε, θα ξέρετε ότι αυτό το καλοκαίρι στη χώρα μου ε, σκοτ, ε, ε, θανατώθηκαν ε, τρεις, τρεις, τρεις αστυνομικοί και έγινε και μια αιματηρή τρομοκρατική επίθεση στην πόλη μου. Θέλω να πω ότι εξακολουθεί για εμάς τους Ισπανούς να είναι πολύ ενισχυτικό το φαινόμενο αυτό. Θα ήθελα να σα ρωτήσω λοιπόν, σκέφτεστε να προωθήσετε νομοθεσία που να προβαίνει σε εναρμόνιση τη ελληνική νομοθεσία, γιατί σήμερα υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά σε θέματα αρρωγή, όχι μόνο οικονομική φύσεω, αλλά και ηθική ε, συνδρομή ε, των θυμάτων ε, τρομοκρατία. Τι θα μπορούσατε να κάνετε εσείς από, από δικού σας οργανισμού. Κατά τα άλλα σα υποστηρίζω και η πολιτική μας ομάδα αλλά και όλοι οι Ισπανοί σας ενθαρρύνουμε να ξεκολουθήσετε να ασκείτε τα καθήκοντά σας με τον τρόπο αυτό. Ευχαριστώ κυρία Λούτφορντ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν να ρωτήσω αν ο κύριος Ντεκέρχοφ έχει ασχοληθεί ποτέ με το θέμα της αποζημίωσης θυμάτων, δηλαδή για πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι θύματα τρομοκρατίας στο εξωτερικό, εκτός της χώρας τους και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο ακόμη δεν το έχουμε επιλύσει αυτό το ζήτημα. Βρετανοί πολίτες δηλαδή, παραδείγματος χάρη, τα θύματα της βομβιστικής επίθεσης στον Παλί, δεν καλύπτονται από κάποιο εθνικό πρόγραμμα αποζημιώσεων. Νομίζω ότι δεν έχει λυθεί ακόμη αυτό το θέμα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και θα ήθελα να ρωτήσω αν γνωρίζετε ποια είναι η κατάσταση και στα άλλα κράτη-μέλη και αν γίνεται κάποια προσπάθεια να βρεθεί μια λύση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεύτερον, συμφωνώ κατά πολύ με τον κύριο Μωράε για το θέμα της έρευνας υπόπτων και στο Ηνωμένο Βασίλειο κάναμε πρόσφατα μια συζήτηση ε, και εδώ λίγο πριν κάναμε μια συζήτηση λίγο πριν έρθετε εσείς σε αυτήν την αίθουσα και συζητήθηκε το θέμα των ε, ε, στοιχείων επιβατών του PNR και η Σουηδική Προεδρία είπε ότι συνεχίζεται το σύστημα των εθνικών συστημάτων PNR και αναφέρθηκε ότι το 80% των κατασχέσεων ναρκωτικών σε ένα αεροδρόμιο της Σουηδίας, νομίζω στη Στοκχόλμη, ε, γίνεται με βάση τα στοιχεία από το σύστημα PNR. Φαντάζομαι ότι αυτό σημαίνει σε μεγάλο βαθμό στοιχεία από την έρευνα υπόπτων. Εξετάζετε λοιπόν εσείς ε, τη χρήση του profiling των ε, στοιχείων που οδηγούν σε έρευνες υπόπτων σε εθνικό επίπεδο και τι επιπτώσεις μπορεί να έχει αυτό στο, σε όλο τον τομέα των ποινικών υποθέσεων. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω ακόμη κάτι που σας είχαμε ρωτήσει και το Σεπτέμβριο, αν έχετε κάτι νέο για τις διατλαντικές σχέσεις σε σχέση με την καταπολέμηση της ε, τρομοκρατίας και το κράτος δικαίου. Έχετε να μας προσθέσετε κάτι σε σχέση με αυτά τα οποία είπαμε το Σεπτέμβριο. Ευχαριστώ, κυρία Αλφάνα. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ήθελα να ρωτήσω την κυρία, τον κύριο Κέρκοφ το εξής. Και είμαι καινούρια ε, στο Κοινοβούλιο και είμαι και εισηγήτρια για το δίκτυο πρόληψη των ε, αδικημάτων, των εγκλημάτων. Ε, λαμβάνοντα υπόψη το πώ έρχονται οι πληροφορίε για την τρομοκρατία και κυρίω το κατά πόσο υπάρχει και πραγματικό feedback απέναντι στις πληροφορίε αυτέ που παρέχονται και το τι γίνεται στη συνέχεια. Και λαμβάνοντα υπόψη ότι ότι απλώνει σε μεγάλο βαθμό τα πλοκάμια, του, τα πλοκάμια της τρομοκρατία ε, και ε, ε επιδίδεται και σε λαθρεμπόριο όπλων και σε εμπόριο ανθρώπων. Αυτό το οποίο θα ήθελα να μάθω και επειδή είμαι συγκήτρια για το δίκτυο πρόληψης ε, των εγκλημάτων είναι ακριβώς να μας πείτε με ποιο μηχανισμό εσείς συλλέγετε πληροφορίες και στη συνέχεια να μας πείτε κατά πόσον οι πληροφορίες που λαμβάνετε επιβεβαιώνονται και από την πραγματικότητα ή και σε στάδιο πρόληψης ευχαριστω κυριε Κύριε Κλέης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κάποια κράτη-μέλη ήδη μίλησαν για την υποδοχή ατόμων από τον Γκουαντάναμο. Άτομα που ήταν ύποπτα συμμετοχή σε τρομοκρατικές δράσεις, χωρίς να υπάρχουν όμως αποδείξεις εναντίον τους. Δεν κατέστη δυνατόν να αποδειχθεί ότι όντως είχαν εμπλακεί σε τέτοιες τρομοκρατικές δραστηριότητες. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε κατά πόσο θα υπάρξει συντονισμός αυτού του θέματος δηλαδή αυτά τα άτομα από τον Γκουαντάναμο που θα κατανεμηθούν σε διάφορα κράτη-μέλη θα έχουν τη δυνατότητα δημιουργίας δικτύων, θα μπορούν να συμμετέχουν σε πολιτικές δραστηριότητες χωρίς όρια, θα ελέγχονται από τις αστυνομικές υπηρεσίες των κρατών μελών. Τι θα γίνει, θα υπάρξει συντονισμός για την παρουσία αυτών των ατόμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Και τώρα κυρία Ντεκέρχοφ θα ήθελα να σας κάνω και εγώ άλλη μια ερώτηση. Μετά τη Λισαβόνα προβλέπεται ότι θα δημιουργηθεί μια νέα επιτροπή εσωτερικής ασφαλείας και θα ήθελα να σας πω, ε, να σας ρωτήσω τι σχέση θα έχει αυτή η Επιτροπή με τη δική σας υπηρεσία συντονισμού αντιτρομοκρατικών δράσεων. Ευχαριστώ πολύ και σας ευχαριστώ για τις εξαιρετικές ερωτήσεις που μου κάνατε. Ακριβέστατες ερωτήσεις και θα προσπαθήσω να τις απαντήσω με τη σειρά που ετέθησαν. Καταρχήν, από τον κύριο Γιώργη Ατόντο για τη συμμετοχή των, υπηρεσιών, των αστυνομικών υπηρεσιών και την ανταλλαγή πληροφοριών. Προσπαθώ κάθε έξι μήνες να υποβάλουμε έκθεση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για διάφορα θέματα τα οποία επιλέγουμε κάπως αυθαίρετα, επιλέγω εγώ τα θέματα που θεωρώ περισσότερο σημαντικά και το θέμα στο οποίο επανερχόμεθα κάθε έξι μήνες είναι ακριβώς αυτό το θέμα, δηλαδή κατά πόσο τα κράτη-μέλη όντως ε, ε, πληρούν το ρόλο τους. Όσον αφορά την ε, Ευρωπόλ και την Eurojust, είναι ο μόνος τομέας για τον οποίο υπάρχει υποχρέωση για τα κράτη-μέλη και βελτιώνονται τα πράγματα. Θα ήταν ε, υπερβολή να πω ότι είναι τέλεια τα πάντα. Ιδίω όσον αφορά την ε, Europol και τι ε, τρέχουσε πληροφορίε, τι έρευνε που είναι ανοιχτέ. Ζωντανέ έρευνε θα τι αποκαλούσα. Κυρίω μεταβιβάζονται στη Europol οι πληροφορίε μετά τι έρευνε. Και εγώ συνεχώ προσπαθώ να εξηγώ στα κρατημέλη ότι είναι απαραίτητο να πληροφορούν συστηματικά την Europol για τι έρευνε που διεξάγονται, που βρίσκονται σε εξέλιξη. Ίσως να πρέπει να τροποποιηθεί κάπως η σχετική νομοθεσία για αυτό το θέμα, δηλαδή ότι υποχρεώνουν τα κράτη-μέλη να ενημερώνουν την Europol μόνο εάν αφορά το θέμα δύο κράτη-μέλη. Και στην αρχή μια έρευνα, είναι δύσκολο να προβλέψει κανεί αν θα υπάρξει κάποια ε, διεθνή εμπλοκή. Όταν υπάρχει λοιπόν διεθνέ θέμα, σοβαρό θέμα, θα είναι σκόπιμο να πληροφορείται η Europol νωρίτερα. Γιατί η Eurojust πρέπει να πούμε ότι ε, στα θέματα τρομοκρατία αργούν κάπω τα και οι πληροφορίε με συστηματικό τρόπο, διότι δεδομένου του ευαίσθητου χαρακτήρα αυτών των στοιχείων, ε, η εκτίμηση είναι ότι συχνά είναι επικίνδυνο να κυκλοφορούν πληροφορίες για μια επικείμενη έρευνα. Διότι αντίθετα με άλλες μορφές τρομοκρατίας, είναι πολύ χρήσιμο να επεμβαίνει κανείς πολύ νωρίς στη διαδικασία για να αποτρέπει οποιαδήποτε ε, ε, επίθεση. Κάτι άλλο στο οποίο προσπαθώ να πείσω τα κράτη-μέλη, είναι δύσκολο και πρέπει ακόμη να γίνει πολλή δουλειά, είναι το να συνεργαστούν η Europol και η Eurojust με τις κοινέ ομάδες ερευνών. Ήμουν στην Europol ε, τις προάλλες με τα 27 κράτη-μέλη για να εορτάσουμε την 10η επέτειο και άκουσα με μεγάλη χαρά πολλούς υπουργούς να λένε ότι επιθυμούν μεγαλύτερη συνεργασία, περισσότερες ε, ομάδες έρευνα και μεγαλύτερη συνεργασία με την Europol και την Eurojust. Και πιστεύω ότι ε, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτά όσον αφορά την αστυνομική συνεργασία. Όσον αφορά τώρα τη συμμετοχή κρατών μελών στην διαμόρφωση πολιτικών, έχω έντονη συνεργασία από τα κράτη-μέλη για ορισμένες στρατηγικές στις οποίες δραστηριοποιούμεθα, ιδιαίτερα σε θέματα πρόληψης και θα σας πω περισσότερα σε λίγο, πολλά κράτη-μέλη δέχτηκαν να συμμετάσχουν, να δεσμευθούν με εμπειρογνωμοσύνη και με πόρους για να προχωρήσουν αυτά τα θέματα και προσπαθούν ε, να κάνουν και ανταλλαγή βελτίστων πρακτικών. Και εδώ θέλω να πω ότι είμαι αρκετά ικανοποιημένο από το δυναμισμό που έχουν δείξει τα κράτη-μέλη. Ένα θέμα στο οποίο επίσης όλα τα κράτη-μέλη κάνουν πρόοδο είναι η δημιουργία μιας πλατφόρμας σε κάθε κράτος μέλος ε, ονομάζεται από πολλούς Fusion Center μέσα στην οποία όλες οι υπηρεσίες όπως ε, υπηρεσίες πληροφοριών, τελωνία, εισαγγελία κλπ. Ε, μοιράζονται τα στοιχεία που έχουν για θέματα τρομοκρατίας. Τα περισσότερα κράτη-μέλη έχουν λίγο πολύ μια παρόμοια πλατφόρμα και υπάρχουν και κάποια κράτη-μέλη που το συζητούν και ένα πρόγραμμα που κάνουμε με την Ισπανία και τη Γαλλία είναι το να δικτυώσουμε αυτές τις πλατφόρμες γιατί κατά αυτόν τον τρόπο θα έχουμε καλύτερη ροή πληροφοριών μεταξύ κρατών μελών. Αυτά για την πρώτη σας ερώτηση. Για τη δεύτερη ερώτηση για την ΕΤΑ ε, δεν υπάρχει αμφιβολία, γι' αυτό την έχουμε και στον κατάλογο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για τρομοκρατική οργάνωση και έχετε δίκιο, πρέπει να χρησιμοποιούμε τις, τους σωστούς όρους και πρέπει να χαρακτηρίζεται ως τρομοκρατική οργάνωση η ΕΤΑ και η συμβασιολογική απόχρωση είναι σημαντική θα έρθω σε επαφή με το Γενικό Διευθυντή Πληροφοριών της ε, ε, Επιτροπής, γιατί δεν το έχουμε συζητήσει, αλλά συμφωνώ μαζί σας ότι η σημασιολογική προσέγγιση είναι σημαντική. Τώρα, στην ερώτηση του κυρίου Μωράες ε, για την έρευνα υπόπτων με βάση θρησκευτική ή εθνοτική ομάδα, και η κυρία Λάτφορντ νομίζω για το ίδιο θέμα επεκτάθηκε. Όντω είναι κάτι που με ανησυχεί και είναι ένα ερώτημα ε, κέρια σημασία. Σε δύο εβδομάδες θα επισκεφθούμε ε, τον οργανισμό που είχατε νομίζω την ε, δυνατότητα να συναντήσετε το διευθυντή του. Υπάρχει Μεγαλο βαθμό διακριτική μεταχείρισης έναντι των μουσουλμάνων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα ήθελα να μπορέσουμε από κοινού να συζητήσουμε αυτά τα θέματα σχετικά με τους συστηματικούς ελέγχους έναντι αυτού που αποκαλούν οι Καναδοί ορατή μειονότητα, πράγμα το οποίο είναι απαράδεκτο. Από ό,τι μου έχουν πει, και ξέρω ότι είναι κάτι που ίσως δημιουργήσει αντιδράσεις, και είναι παράδοξο για αυτούς που είναι κατά του PNR, μου λένε ότι το PNR αποφεύγει ακριβώς αυτούς τους ελέγχους που βασίζονται σε εμφανείς ορατές μειονότητες. Πάντω έχετε δίκιο για αυτή την ερώτηση και έχω δει και κάποιε μελέτε ε, και απαιτείται και περαιτέρω εργασία και είναι κάτι που πρέπει να μα απασχολήσει από κοινού με το Συμβούλιο. Τώρα επανέρχομαι στην ερώτησή σα για την πρόληψη. Αυτό ήταν άμεση η προτεραιότητά μου όταν διορίστηκα, διότι νομίζω ότι πρέπει να καταβάλουμε μεγάλες προσπάθειες από αυτού. Η δυσκολία είναι ότι κυρίως είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών. Και θα πρέπει να πείσουμε τα κράτη-μέλη να επενδύσουν, να μοιράζονται τις πρακτικές τους και να κάνουν ανταλλαγή βελτίστων πρακτικών. Μέχρι τώρα έχω καταφέρει να βρω έξι πρόθυμα κράτη-μέλη που να θέλουν να συμμετάσχουν ε, σε αυτό το προληπτικό πρόγραμμα για θρησκευτικού ηγέτε, για το πώ μπορούμε να αναπτύξουμε ε, μια πολιτική αντιστροφή των τάσεων και πώς μπορούμε να κινητοποιήσουμε τους, ανθρώπου ανθρώπους σε τοπικό επίπεδο, γιατί σε τοπικό επίπεδο πρέπει να κινητοποιήσουμε οικογένειες, ε, κοινωνικού κοινωνικούς λειτουργούς, σχολεία κλπ. Επίσης προσπαθούμε ε, να δουλέψουμε πάνω στην ε, ελάττωση των ριζοσπαστικών τάσεων. Με ένα κράτος μέλος ήδη το κάνουμε αυτό. Και σας ομολογώ ότι είναι μεταξύ των ε, κυρίων προτεραιοτήτων μου. Είναι πολύπλοκο το θέμα και όσο πιο πολλά διαβάζω τόσο λιγότερα αντιλαμβάνομαι ότι γνωρίζω και οποιαδήποτε συνεισφορά σας θα είναι ευπρόσδεκτη. Όσον αφορά τώρα την ερώτηση της Σοφίντφελντ για την πρόσφατη ε, απόφαση του δικαστηρίου, νομίζω ότι θα πρέπει να χαιρόμαστε που έχουμε το δικαστήριο. Γιατί το δικαστήριο μας βοηθάει να επαναρθώνουμε σφάλματα. Όπως και εσείς, δεν θα ήμουν τόσο αρνητικός ως προς την αλλαγή διαδικασίας Πρέπει να βελτιώσουμε τη διαδικασία blacklisting μετά από κάποιες αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Θέλουμε να υπάρχει μια δίκαιη διαδικασία και δεν έχω δει καμία καινούργια απόφαση του δικαστηρίου ή του πρωτοδικίου που να αμφισβητεί τη νέα διαδικασία που έχουμε εγκαθιδρύσει Το ΣΑΙΖΟ ή το ΚΟΖΙ δεν είναι επιχείρημα για να αλλάξει η διαδικασία, αλλά το, το ότι μπήκε στο κατάλογο στην Ολλανδία αυτή η οργάνωση είναι γιατί δεν τους δόθηκε η δυνατότητα να αμφισβητήσουν, να ασκήσουν ένσταση για την ε, συμπερίληψή τους στον ε, κατάλογο, στο blacklist. Νομίζω λοιπόν ότι είμαι βέβαιο ότι η διαδικασία έχει βελτιωθεί σημαντικά. Αλλά όσο περισσότερο μπορούμε να βελτιώνουμε τι διαδικασίε, τόσο το καλύτερο. Και από τη νέα συνθήκη ένα ιδιαίτερα θετικό σημείο είναι ότι θα μα επιτρέψει τη δημιουργία ενό μηχανισμού για την τρομοκρατία και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Και όταν υποβάλει η πρόταση η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο θα συνεργαστεί και ελπίζω ότι θα καταλήξουμε σε μια θέση που θα πληρεί όλες τις απαιτήσει σας. για την πιο εμπεριστατωμένη πολιτική, νομίζω ότι ήδη έχω απαντήσει σε αυτήν την ερώτηση, είναι κάτι που πολλές φορές λείπει και στο πλαίσιο της νέας συνθήκης η αξιολόγηση είναι ένας μηχανισμός στον οποίο επιμένει η νέα συνθήκη και θα σχεδιάσουμε ένα μηχανισμό αξιολόγησης μετά από λίγα χρόνια για να είναι σίγουρο ότι έχουμε το σωστό όργανο στη διάθεσή μας, όχι μόνο για την νομική εφαρμογή αλλά και για το αν είναι δίκαιο και αποτελεσματικό το σύστημα. Για το Ισλάμ και τους μουσουλμάνους, και εγώ προσπαθώ να μην εστιάζουμε ε, με ασφαλμένο τρόπο, να μην χρησιμοποιούμε ατυχείς όρους, και να μην χρησιμοποιείτε, να μην εκμεταλλευόμαστε τη θρησκεία για πολιτικούς ε, λόγους, όταν δεν υπάρχει κανένας λόγος να αναφέρει τη θρησκεία, επομένω συμφωνώ μαζί σας. Και χάρη στις υπηρεσίες ε, πληροφοριών και ασφαλείας και το DSAT δεν έχει ε, δημιουργήσει κανένα αρνητικό καμιά αρνητική εξέλιξη και δεν είχαμε και καμιά ε, τρομοκρατική επίθεση σε μεγάλο βαθμό μετά από αυτές στο Λονδίνο. Πρέπει να πούμε ότι με διμερείς συνεργασία μεταξύ Γαλλίας και Ισπανίας ε, ε, ε, δόθηκε κάποια απάντηση στο πρόβλημα της ΕΤΑ και πολλά μπορούμε να πούμε για την διμερή συνεργασία και θα ήθελα να πω ότι είναι σωστή απάντηση η αντιτρομοκρατική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν δαπανούμε πόρους σε κάτι το άσχετο. Και θα ήθελα να απαντήσω και στην κυρία Βεσέιλ. σχετικά με τον ορισμό της τρομοκρατίας. Υπάρχει ένας ορισμός της τρομοκρατίας από το 2002, ο οποίος διευκρινίστηκε κάπως το 2008 και καλύπτει και άλλες συμπεριφορές όπως ε, την προτροπή προς διάπραξη εγκληματικής πράξης. Αλλά όντως ε, πρέπει ο ορισμός να διατυπώνεται σωστά και να ανταποκρίνεται στην εξέλιξη του φαινομένου. Γι' αυτό το 2008 τροποποιήσαμε τον ορισμό του 2002, ώστε να λάβουμε υπόψη μας και νέες συμπεριφορές που είχαν παρατηρηθεί ως τότε. Μια ερώτηση είναι το αν θα ήταν χρήσιμο, διότι είναι ένα φαινόμενο που παρατηρείται από τις υπηρεσίες πληροφοριών, αν θα ήταν ε, σκόπιμο να ποινικοποιήσουμε την μετάβαση σε μια άλλη χώρα για να ε, συμμετάσχει κανείς σε κάποιο στρατόπεδο εκπαίδευσης, όπως το Πακιστάν παραδείγματος χάρη. Είναι μια ερώτηση αυτή. Ξέρω λοιπόν ότι ε, πρέπει να σας πω ότι έχουμε έναν ορισμό για τον οποίο υπάρχουν ενστάσεις από πολλούς, αλλά νομίζω ότι είναι σωστός ο ορισμός και θα πρέπει να συνεχίσουμε να παρακολουθούμε την εξέλιξη των όρων. Ε, όσον αφορά την έκδοση τρομοκρατών. Θυμάμαι κάποιο κράτο μέλο που γνωρίζω πάρα πολύ καλά που δεν ε, που αρνείται να εκδώσει προ την Ισπανία ε, μέλη τη ΕΤΑ και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν είναι πλέον δυνατόν διότι έχει αλλάξει η κατάσταση με το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψη. Εξαρτάται βέβαια και από τη διαδικασία που υπάρχει για τη σύναψη συμφωνιών ε, έκδοσης και εδώ ακριβώς μια ισχυρή πολιτική Ευρώπη θα πρέπει να είναι σε θέση να κάνει μια τέτοια συζήτηση και να καταλήγει σε μια τέτοια ε, συνθήκη και μέσα στα επόμενα χρόνια θα πρέπει οι υπουργοί μας να έρθουν σε επαφή με τις γειτονικές χώρες με όσους είναι υπεύθυνοι για το λαθρεμπόριο ναρκωτικών ή για την τρομοκρατία και να συνάψουν τέτοιες συμφωνίες. Ήμουν το καλοκαίρι στην Κολομβία και για θέματα έκδοσης θα μπορούσαμε να σκεφτούμε τη δημιουργία μιας τέτοιας συμφωνίας με την Κολομβία για την έκδοση εμπόρων ναρκωτικών όπως έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Για την ερώτηση της κυρίας Λάτφορντ, πρέπει να αφιερωθούμε περισσότερο στο θέμα της αποζημίωσης των θυμάτων. Δεν μπορώ να σας πω λεπτομέρειες για το αν καλύπτονται τα θύματα στο εξωτερικό από τις ασφαλιστικές εταιρείες κλπ. Νομίζω πως όχι και όντως είναι κάτι το οποίο πρέπει να διερευνήσουμε και θα προσπαθήσω να το ερευνήσω και να σα δώσω μια πιο συγκεκριμένη απάντηση. Και για την τελευταία σχέση, για την τελευταία ερώτηση, συγγνώμη, για τη σχέση με του Αμερικανού. Νομίζω ότι είπα και την προηγούμενη φορά στην κοινή δήλωση Ευρωπαϊκή Ένωση ΗΠΑ για τον Γκουαντάναμο είχε συμφωνηθεί να αρχίσει μια διαπραγμάτευση αρχό, κοινών αρχών για την καταπολέμηση τη τρομοκρατία. Και ε, ε, στην κοινή δήλωση και στα συμπεράσματα του Συμβουλίου είπαμε, πράγμα που είπα και σε πρόσφατες συνεντεύξει, ότι αυτό το κάναμε θεωρώντας ότι οι Αμερικανοί θα άλλαζαν το μοντέλο τους και θα περνούσαν σε ένα άλλο μοντέλο εφαρμογή της νομοθεσίας. Γίνεται συζήτηση τώρα σχετικά με το θέμα αυτό και στην Ουάσιγκτον και είναι δύσκολο να σας δώσω κάποια αποτελέσματα γιατί ανεβλήθη η υποβολή της τελικής έκθεσης από την Task Force που χειρίζεται με το θέμα. Αλλά πάντως ε, ε, εργαζόμαστε πάνω σε αυτό το θέμα. Και είμαι σε επαφή με το νομικό σύμβουλο του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ και τον συντονιστή κατά της τρομοκρατίας του Υπουργείου Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών για να δούμε πώς μπορούμε να προχωρήσουμε. Θα ξεκινήσει νομίζω όμως με την επερχόμενη Ισπανική Προεδρία γιατί θέλουν οι Αμερικανοί να περιμένουν την έκθεση για την πολιτική κράτησης. είναι ένα από τα θέματα που έχω στην ημερήσια διάταξη για τη συνάντηση που θα κάνουμε με τον Αμερικανό Αντιπρόεδρο στην Ουάσιγκτον στα τέλη Οκτωβρίου. Θα πιέσω για αυτό το θέμα. Για την ερώτηση τη κυρία Αλφάνο, εμπόριο όπλων και εμπόριο ανθρώπων, αν έχουμε επαρκεί πληροφορίες. Τα τελευταία χρόνια νομίζω ότι έχουν ε, βελτιωθεί πάρα πολύ οι πληροφορίες της ε, Europol και έχουμε όλο και πιο λεπτές αναλύσεις και υπάρχει το CITSEN, το κέντρο ε, το οποίο διαχειρίζεται αυτά τα θέματα και νομίζω ότι και τα Υπουργεία Δικαιοσύνη και Οικονομικών έχουν πολύ πιο ευαίσθητε πληροφορίες, ε, πληροφορίες που τους επιτρέπουν να καθορίσουν πιο σωστά την πολιτική που θα ακολουθήσουν. Όσον αφορά το Γκουαντάναμο, όπως γνωρίζετε, τον Ιούνιο το Συμβούλιο ΔΕΗ ενέκρινε ένα μηχανισμό που επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών για τα κράτη-μέλη που έχουν κατά νου ε, να υποδεχθούν έναν ή περισσότερους κρατουμένους και στη συνέχεια, στο πλαίσιο των αρχών του Συμβουλίου, προβλέπεται η ανταλλαγή πληροφοριών για το καθεστώς, για τον τρόπο με τον οποίο γίνεται αποδεκτά στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτά τα άτομα. Κράτη-μέλη ε, τα οποία υποδέχονται ε, κρατουμένους θα πρέπει να σέβονται τις ευαισθησίες άλλων κρατών μελών. Ένα κράτος μέλος θα πρέπει να πληροφορεί τα άλλα κράτη-μέλη για ενδεχόμενα μέτρα ασφαλείας. Ίσως να πρέπει ε, να αναφέρεται στην αστυνομία κάθε εβδομάδα ή θα πρέπει να παρακολουθείτε από κάποιες μυστικές υπηρεσίες, αλλά θα πρέπει να ενημερώνει το κάθε κράτος μέλος τα άλλα κράτη-μέλη. Νομίζω ότι οι σχετικοί μηχανισμοί λειτουργούν σωστά πληροφορούν τα κράτη-μέλη το ένα το άλλο για τα μέτρα τα οποία λαμβάνουν και θα προσπαθήσουμε να τηρήσουμε και τα νομικά μέτρα σχετικά με το καθεστώς αυτών των ατόμων, αλλά και τα μέτρα τα οποία επιβάλλονται για την ένταξή τους, γιατί είναι σημαντικό να εξασφαλίσουμε την σωστή ένταξη αυτών των ατόμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για, το ρόλο του, για την ερώτηση του Προέδρου σχετικά με το ΚΟΖΙ και το ρόλο που θα μπορούσαμε να έχουμε εμείς. Το ΚΟΖΙ θα είναι ε, κάτι δύσκολο αλλά πολύ σημαντικό. Θα είναι δύσκολο διότι μέχρι τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση ποτέ δεν κατάφερε, δεν κατάφερε όσον αφορά την εσωτερική ασφάλεια να αναπτύξει την ε, λειτουργική συνεργασία. Ε, κάνουμε ε, επιχειρησιακή συνεργασία 27 ε, κρατών μελών και είναι δύσκολο να το κάνουμε στην Europol. Είναι τεράστια η πρόκληση και θα πρέπει όλοι οι εταίροι να συνεργαστούν. Η Europol, η Eurojust, η Olaf, η Frontex θα πρέπει να συνεργαστούν για να δούμε ποιε είναι οι προτεραιότητε μιας πολιτικής κατά της τρομοκρατίας. Είναι ένα από τα θέματα με τα οποία θα ασχολείται το ΚΟΖΗ. Τα κράτη-μέλη προσπαθούν, προτιμούν να έχουν κάποιο πολυμερές σύστημα ανταλλαγή πληροφοριών, αλλά νομίζω ότι το ΚΟΖΗ θα έχει να παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο και για εξοικονόμηση πόρων. Και θα χρειαστεί βέβαια κάποιος χρόνος μέχρι να βρει το ρυθμό του το ΚΟΖΗ, Αλλά μετά από 10 χρόνια λειτουργίας της Europol, βλέποντας τις βελτιώσεις που έχουν επέλθει, είμαι αισιόδοξο για το πλαίσιο αναφοράς στο οποίο θα καταλήξουμε και σε αυτό το τομέα. Με το πρόγραμμα COSPOL, με το ΟΚΤΑ, προσπαθήσαμε ε, να ε, εξετάσουμε πεδία πολιτικής για ποινικές ε, υποθέσεις και τον ίδιο τρόπο θα πρέπει να διασφαλίσουμε να συνεργάζονται όλες οι υπηρεσίες στα κράτη-μέλη. Το άρθρο λοιπόν για το κόζι λέει ότι, δεν το έχω μπροστά μου βέβαια, πάντως λέει ότι όλοι όσοι έχουν σχέσεις Μισό λεπτάκι να το βρω για να σας το διαβάσω. Οι εκπρόσωποι των ε, οργάνων και οργανισμών που θα συνεργάζονται για αυτά τα θέματα. Τώρα βέβαια εμείς δεν ξέρω αν είμαστε όργανο ή οργανισμός. Πάντως και ο συντονιστής θα έχει κάποια θέση στο πλαίσιο του ΚΟΖΗ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ζιντεκερκόφ. Ε, γνωρίζουμε ότι είστε συντονιστής ε, του προγράμματος ε, δράσης για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, συντονιστής των αντιτρομοκρατικών ενεργειών. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα αυτά που μας είπατε. Θέλει κανείς άλλος να πάρει το λόγο ο κύριος Μπρόνς, ε, κοιτάξτε, δράτω με της ευκαιρίας να ζητήσω αλλά την αντικατάστασή μου στην Προεδρία. Μπορείς να έρθει σε παρακαλώ ε, να έρθει η κυρία Ίντβελτ ε, γιατί πρέπει οπωσδήποτε να φύγω. Η κυρία Ίντβελτ λοιπόν θα πάρει τη θέση μου στην Προεδρία. Safe trip home. Uh, Mrs. Hennis. Η κυρία Ευχαριστώ. Μία ερώτηση πάρα πολύ σύντομη, γιατί και εγώ δυστυχώς πρέπει να φύγω. Στις 6 ακριβώς ε, το αργότερο. Ε, νομίζω, όπως κατάλαβα, ότι υπάρχει νέα συμφωνία με, τα, με τις Ηνωμένε Πολιτείες. Και επομένως το ερώτημά μου είναι το εξής. Ε, αυτό σημαίνει βάσει τη νέα συμφωνία ότι θα πρέπει να δώσουμε ε, τα δεδομένα μα στι Ηνωμένε Πολιτείε. Ε, δεδομένα τα οποία οι Ηνωμένε Πολιτείε θα αναλύσουν και επομένω θα φαντάζομαι ότι θα έχουμε και ροή πληροφοριών από τις Ηνωμένες Πολιτείες προς εμάς. πρόκειται για στοιχεία τα οποία είναι απολύτως απαραίτητα φαντάζομαι για την αντιτρομοκρατική γιατί, γιατί τελικά όμως, και αυτή είναι η ερώτησή μου, γιατί αφήνουμε τους Αμερικανούς να διαχειρίζονται εκείνοι αυτά τα δεδομένα. Από ό,τι βλέπω, λέει η Πρόεδρος, υπάρχει άλλη μία ερώτηση. Μετά από αυτήν θέλει κάποιος, α, και ο κύριος Μπουζουτήλ. Ωραία. Μπρόνς και μετά Μπουζουτήλ. Ευχαριστώ πολύ. Ε, Βεβαίω γνωρίζουμε ότι η Ισλαμική τρομοκρατία δεν είναι η μόνη τρομοκρατία. Αλλά σε σχέση με αυτήν την ειδική μορφή τρομοκρατίας, ποια θα είναι η σχέση με τις ε, μουσουλμανικές ε, χώρες, το Ιράκ και ενδεχομένως το μέλλον του Ιράκ και κατά πόσον μπορούμε να θεωρήσουμε ότι υποθάλπτουν τρομοκρατίε και τρομοκρατικέ ενέργειε. Ο κύριος Μπουσουτήλ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Μια πολύ απλή ερώτηση. Έχετε, κάνει κάποια διασύνδεση ανάμεσα στην παράτυπη ή λαθρέα μετανάστευση και την ε, ε, τρομοκρατία. Ξέρουμε ότι υπάρχει μεγάλη μετακίνηση από τη Βόρεια Αφρική προς ε, την νότια παράλια της Ευρώπης. Υπάρχει κάποια διασύνδεση, κύριε Δικερκόφ. Ναι όσον αφορά την πρώτη ερώτηση, φαντάζομαι ότι σχετίζεται με το SWIFT. Ε, ναι, είχα ξανά την ε, ευκαιρία να ξαναμιλήσω για το πρόγραμμα ανίχνευσης τρομοκρατών, ε, το οικονομικό αυτό πρόγραμμα. Ε, πρέπει να σας πω ότι πρόκειται για μια πρόσκαιρη συμφωνία με χρόνο ε, ζωής το ένα έτος. Αλλά όσον αφορά το συγκεκριμένο σας ερώτημα, ε, λαμβάνοντας υπόψη είναι μια αλλαγή στο οικοδόμημα, στην αρχιτεκτονική του οικοδομήματος, είναι ε, γεγονός ότι υπήρξαν κάποιες αλλαγές. Εγώ δεν λέω ότι το σύστημα δεν είναι σωστό, όμως συμφωνώ μαζί σας ότι θα πρέπει να αποφασίσουμε ποιο θα, ποιο θα είναι το μέλλον αυτού του μηχανισμού και επομένως θα πρέπει να δούμε κατά πόσον πρέπει να έχουμε το UTFTP. η παρούσα ε, συμφωνία και θα δούμε αν βεβαίως συμφωνηθεί τελικά από τους ε, υπουργούς ε, σημαίνει ότι θα μπορούσαμε να έχουμε σε μια μέρα ένα νέο UTFTP. Όσον αφορά το Ιράν και το Ιράκ, δεν θέλω να σχολιάσω για το Ιράκ, γιατί τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά, το ξέρουν όλοι. Έχουμε μια εξωτερική πολιτική η οποία προωθεί τις ε, ε, καλές εξωτερικές σχέσεις, την ε, καλή διακυβέρνηση και βεβαίως την ανεξαρτησία των, και την εθνική κυριαρχία των κρατών, των τρίτων κρατών. Αναφερθήκατε σε μια ατμόσφαιρα και την ατμόσφαιρα του Ιράν. Εγώ δεν θέλω οπωσδήποτε να γίνει αναφορά στο Ιράν, αλλά νομίζω ότι πραγματικά υπάρχουν πολλά θέματα που διακυβεύονται εδώ και τα οποία είναι πάρα πολύ σοβαρά. Φυσικά μας ενδιαφέρει η χώρα όχι μονάχα μεμονωμένα αλλά και σαν παράγοντα σταθερότητας. Όσον αφορά τη διασύνδεση ανάμεσα στη μετανάστευση και, και την τρομοκρατία δεν βρίσκουμε καμία διασύνδεση. Ε, υπάρχουν μορφές ε, γηγενούς ε, τρομοκρατικής δράσης στην Ευρώπη που δεν έχει καμία σχέση με την μετανάστευση ξέρουμε ότι σε πολλές περιπτώσεις έχουμε ελέγξει χρόνο, τρόπο συγγνώμη, προετοιμασίας τρομοκρατικών δράσεων που δεν έχει καμία σχέση με την μετανάστευση. βεβαίως Βεβαίως ξέρουμε ότι στην περίπτωση της επίθεσης 10 Σεπτεμβρίου υπήρχαν άτομα τα οποία έφτασαν πρώτα στην Ευρώπη και μετά από την Ευρώπη πέρασαν στις ΗΠΑ. Πολιτείες και γι' αυτό θεωρούμε ότι είναι σημαντικός και ο έλεγχος στα σύνορα. Είναι σημαντικό το να συλλέγουμε πληροφορίες. Είναι σημαντικό να δούμε κατά πόσον μπορούμε να απομονώσουμε τους τρομοκράτες ε, την στιγμή που ταξιδεύουν ή τη στιγμή που περνούν τα σύνορα. Αλλά ακριβώς εδώ υπάρχει και ο κίνδυνος του να, να μπερδέψουμε διαφορετικά πράγματα, δηλαδή το έγκλημα, την τρομοκρατία και την μετανάστευση. Θα πρέπει οπωσδήποτε να προάγουμε την ασφάλεια των ταξιδιωτών ε, και από την άλλη πλευρά να προάγουμε και την, το σύστημα πληροφοριών που έχουμε όσον αφορά τους ταξιδιώτες, αλλά να μην υπάρξει απαραίτητα διασύνδεση ανάμεσα στην τρομοκρατία και την μετανάστευση. Ευχαριστώ. Αν μου επιτρέπετε να κάνω μια ηρωνική παρατήρηση. Νομίζω ότι πολύ λίγοι είναι οι παράνομοι μετανάστες που περνάνε ε, την ε, Μεσόγειο σε μικρές βάρκες και αυτό το βλέπετε μέσα στα αρχεία PNR. Λοιπόν, ε, όσον αφορά την ερώτηση του συναδέλφου, δεν είχε να κάνει τόσο με το, Ιρα... με το γεγονός ότι το Ιράκ και το Ιράν είναι Ισλαμικές χώρες. Αλλά αν δείτε την ριζοσπαστικοποίηση όπως και το κάνετε, και αν δείτε κάποια ένδειξη ότι αυτοί οι πόλεμοι χρησιμοποιούνται ως πρόσχημα για διεξαγωγή αυτών των δημοκρατικών ενεργειών. Αυτό, αυτό ήταν η ερώτηση. Είχε να κάνει με το αν ακριβώ χρησιμοποιούν ως πρόσχημα το Ισλάμ. Κύριε Μπουσούτη, και να προσθέσετε κάτι, άμα επιτρέπετε. Την επόμενη φορά. Να ξεκαθαρίσω. Δεν είχα του ε, στο μυαλό μου του μετανάστε που έρχονται παράνομα και το γεγονό ότι μπορεί να είναι τρομοκράτε, αλλά τη χρηματοδότηση των εγκληματικών οργανώσεων που βρίσκονται πίσω από το εμπόριο ανθρώπων. Ε, η οποία ε, είναι με ιδιαίτερα δικτυωμένη, η οποία είναι ιδιαίτερα δικτυωμένη αυτοί οι άνθρωποι. Και η ερώτησή μου είναι εξή. Έχετε εξακριβώσει τη συσχέτιση ανάμεσα αυτού του είδου στι εγκληματικέ οργανώσει και στη χρηματοδότηση τη τρομοκρατία. Α, δεν είχα καταλάβει υπάρχουν κάποιες εγκληματικές ομάδες όπως για παράδειγμα το PKK στην Τουρκία που όπως έχει υποδείξει η αστυνομία ε, επιδίδεται σε αυτό το εμπόριο όπλων ε, όχι για επιθέσεις στην ε, τρομοκρατία αλλά στο βόρειο Ιράκ. Ναι, συμβαίνει αυτό, πράγματι. Ναι, μπορεί να συμβεί αυτό που είπατε αλλά δεν έχει να κάνει μόνο με το εμπόριο ανθρώπων και δεν έχει να κάνει μόνο με την μετανάστευση, αλλά συσχετίζεται σε γενικέ γραμμέ με οποιαδήποτε φύση ω Όσον αφορά την πρώτη ερώτηση. Ναι. Ε, αναφέρεται τέτοια χρήση και αν δείτε ε, τον ίδιο τον Οσάμα Μπιν Λάδεν... και τη ρητορική του και το πώς χρησιμοποιεί λανθασμένο για να παραπλανήσει οποιοδήποτε, οποιοδήποτε γεγονός σε διεθνές επίπεδο και οποιοδήποτε εκδήλωση για να τροφοδοτήσει τα δικά του επιχειρήματα. Η ακουσία λύσεως στη Μέση Ανατολή είναι το διαρκές του επιχείρημα. Και βεβαίω είναι κάτι που πρέπει να επιληθεί όσο το πιο γρήγορα και που δεν έχει επιληθεί σε συλλογικό επίπεδο μέχρι στιγμή. Ε, και βεβαίω το χρησιμοποιούν ω πρόσχημα. εισβολή στο Ιράκ. Έχει χρησιμεύσει ως πρόσχημα και, ε, ως, και το έχει τροφοδοτήσει τη ρητορική πολλών ομάδων. Ευχαριστούμε. Το τελευταίο αυτό ζήτημα αποδεικνύει ότι αν θέλουμε να φτάσουμε στις καρδιές και στο μυαλό των ανθρώπων, πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι εμείς διατηρούμε ε, το δικό μας ηθικό κύρος ε, και ότι δεν δίνουμε ε, πρόσχημα σε κανέναν για να επιδοθεί λόγω των πράξεών μας σε τρομοκρατικές δραστηριότητες. Σε ευχαριστούμε. Κοιτάξτε, επίσης τέλος του μήνα θα έχουμε μια αντιπροσωπεία της Επιτροπής μας που θα μεταβεί στις Ηνωμένες Πολιτείες για να συναντηθεί με τους ομολόγους μας στο Κογκρέσο. Μήπως θα μπορούσατε ε, ε, να έρθετε ε, για να κάνουμε μια σύντομη ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων εν ώψη αυτή ακριβώ τη αντιπροσωπεία. Α, θα είστε και εσεί στην Ουάσιγκτον δεν Πάρα πολύ ωραία. Άρα λοιπόν είστε διαθέσιμο για κάποια σύντομη προετοιμασία μαζί μας. Α, αυτή η τελευταία παρατήρηση βλέπω ότι έδωσε έναυσμα στη Σάρα. Και μετά λέω να τελειώσουμε. Προς ενημέρωσή σας το Προεδρείο ε, της Αντιπροσωπείας των Ηνωμένων Πολιτειών θα μεταβεί ταυτόχρονα. Και επειδή είμαι η πρώτη αντιπρόεδρος αυτής της αντιπροσωπείας, νομίζω ότι η ιδέα είναι, παρόλο που δεν έχει αναφερθεί σαφώ, είναι να υπάρξει ε, αυτή η συνεργασία με την Επιτροπή Λίμπα και να είμαι και εγώ με διαφορετικό καπέλο. Άρα σα παρακαλώ, θα ήθελα να με συμπεριλάβετε σε οποιαδήποτε μορφή σε ενημέρωση. Πολύ ωραία, σα ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω και αν κάποιο θέλει να πει κάτι στα διάφορα. Διαφορετικά θεωρούμε ότι έλειξε η συνεδρίασή μα. Ευχαριστώ. Αύριο το πρωί στι 10 από ό,τι μου λένε οι συνάδελφοι. 10 ακριβώ όμω.